Αξιότιμε meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Προσωρινή ημερήσια διάταξη μπορούμε να την κάνουμε δεκτή, αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Όλο το εξαιρετικό συνεδρίαση των συντονιστών θα ξεκινήσει αύριο στι 9 το πρωί για λόγου καθαρά οργανωτικού. Άρα οι ψηφοφορίε αύριο θα γίνουν στις 10. Εάν δεν έχετε αντιρρήσει επίση μπορούν να εγκριθούν τα πρακτικά της 4 η και 5 η Μαΐου. Σήμερα έχουμε δύο ομάδε επισκεπτών. ορίσω καταρχάς θερμά αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, Μεταφορών του Ειδικού Κοινοβουλίου. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ο κύριος Ρικέ έχει προσκαλέσει εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, Εθνικής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών της Πικαρδίας. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Προχωρούμε λοιπόν, για να δείτε και εσείς πώς δουλεύουμε. Επόμενο θέμα της ημέρας της διάταξης, περιορισμός των ρηπογόνων εκπομπών από ε, οχήματα οδικής χρήσης με την κυρία Εσβίατα Λουκασίγεβα στην οποία δίνω και το λόγο αμέσως, που είναι... Εσβίατα Λουκασίγεβα έχετε το λόγο. Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω όλους τους χειόδους ηγητάς θερμά για όλα τα σχόλια που έλαβα από πλευρά σας. Ε, προσπάθησα ε, να τα συμπεριλάβω όλα στην γνωμοδότησή μου. Έχετε λάβει φαντάζομαι την τελική έκδοχη της γνωμοδότησης αυτής και ελπίζω ότι σας ικανοποιεί. Υπενθυμίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο κανονισμούς, έγκριση των ε, κινητήρων για ελαφρά οχήματα, Euro 5 και Euro 6 και αντίστοιχα οχήματα ε, φορτηγά με βαρύ φορτίο, πάλι θέμα περιορισμού των ρηπογόνων εκπομπών. Προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτές τις εκπομπές, αλλά ταυτόχρονα και την ε, επιβάρυνση για τον ε, παραγωγό, για τον κατασκευαστή σε όρους ε, γραφειοκρατίας. Έχουμε μία σειρά από τροπολογίες. Ιδιαίτερο θέμα είχαμε την αύξηση της χρήσης των ε, καυσίμων που εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα. Είχαμε συναδέλφους που θέλαν να αφήσουν σε κατεξουσιοδότηση πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ρύθμιση αυτήν. Άλλοι που θέλαν να διατηρηθεί η συνήθις νομοθετική διαδικασία. Είναι ένα θέμα τεχνικό. Έχουμε δύο συμβαστικέ τροπολογίες για το μεθάνιο αφενός, ύστερα από τι διαβουλεύσει με τι ομάδε αποφασίσαμε να απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, εκπόνηση κανονισμού μετά τις πρώτες συζητήσεις και τη διερεύνηση των θέσεων του κλάδου, των κατασκευαστών και λοιπόν ε, ενδιαφερομένων πλευρών εξετάσαμε πώς μπορεί να επηρεάσει το κείμενο αυτό την κατασκευή και τις εκπομπές, ιδίως για οχήματα που χρησιμοποιούν αέριο. Και καταλήγουμε σε μια απόφαση η οποία σε στόχο έχει ιδιαίτερα να ενθαρρύνει τον καταναλωτή ε, να χρησιμοποιεί περισσότερο οχήματα κινούμενα με αέριο. Επίσης προσπαθούμε να κοιτάξουμε να κάνουμε πιο ελκυστικά, έστω και αν δεν είναι. Ε, να κάνουμε να γίνουν λιγότερο ελκυστικά, όσο και αν δεν είναι σωστό όρο ελκυστικά, αλλά να είναι λιγότερο ελκυστικά τα οχήματα με δίζελ. Χρησιμοποιούν δίζελ. Γιατί θεωρούμε ότι έχουν ε, ιδιαίτερη συμμετοχή στην ε, αύξηση των ρηπογόνων εκπομπών. Εδώ λοιπόν η Επιτροπή ζητεί μια κατεξοδότηση πράξη. Εμείς θα μπορούσαμε και να διαγράψουμε τη σχετική παράγραφο, αυτή που αναφέρεται δηλαδή σε νέα όρια. Εγώ νομίζω ότι εφόσον αυτό δεν επηρεάζει τις εκπομπές καυσαερίων, βλαβερών καυσαερίων, μπορούμε να διαγράψουμε τα ποσά, αλλά όχι ολόκληρη την παράγραφο έχει γίνει συζήτηση με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω λάβει μια σειρά από παρατηρήσεις και σχόλια, στις οποίες προσπαθώ με το κείμενό μου και τις τροπολογίες μου να δώσω απαντήσεις. Μετά τις συζητήσεις με διαφόρους εμπλεκομένους και κατασκευαστές βεβαίως οχημάτων, μπορώ να πω ότι ελπίζω πως οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες θα σας βρουν σύμφωνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ισκιώδη και κυρία Ρεβό. Merci, Président. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για αυτή την συνεργασία που είχαμε. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία το λέω γιατί Μπορεί να καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά μετά ο χαμένος χρόνος κερδίθηκε και τα πήγαμε περίφημα. Για την τεχνική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να καταλάβετε πως οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις εκπομπές αυτές αποτελούν ένα από τους βασικούς άξονες για τη μάχη κατά της ρήπανσης που θίγει τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη καθημερινά. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση αυτή, η οποία ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, αυτή που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει και η έκθεσή μας. Χρειαζόμαστε για το διοξίδιο αζότου κάποια όρια, ανώτατα όρια, ε, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θεσπίσει και που χειροτερεύουν την ε, ρήπανση στο αστικό περιβάλλον. Επίσης, υδρογοναθρακές θα πρέπει να έχουμε εναλλακτικά οχήματα στην αγορά που να χρησιμοποιούν αέριο για να μειώσουμε τη ρήπανση. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Για να βελτιώσουμε την πρόταση θα ήθελα να κάνω τις εξής προτάσεις. Καταρχήν μια σειρά τροπολογιών έτσι ώστε να έχουμε κάποιες δοκιμές που θα γίνονται υπό πραγματικές συνθήκες. Γιατί οι κατασκευαστές θα πρέπει να κάνουμε μια προσωμείωση με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης τη στιγμή που δοκιμάζουν τα οχήματά τους έτσι ώστε να γίνονται σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες, κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι συμβαίνει σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, είναι όμως απαραίτητο να αναφερθούμε στο κείμενο αυτό στις ε, πραγματικές συνθήκες ε, για να το εξασφαλίσουμε. Τώρα, για το πώς υπολογίζουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να σας πω πώς θα πρέπει να δούμε πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις και αν με κάποιο τρόπο μπορούμε να προκρίνουμε τα οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. Για τις εκπομπές υδρογονάνθρακων θα πρέπει ίσως να έχει ένα ισοδύναμο για το διοξείδιο του άνθρωπου μεταξύ μέσω κατεξουσιοδότησης πράξης, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Αυτή η συμπερίληψη του μεθανίου στο του διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να γίνει σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους περιορισμούς της εκπομπές που θα ισχύσει από το 2016. γιατί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζω τις τροπολογίες της εισηγήτριας και νομίζω πως θα πρέπει αυτή την ε, μοιρασμένη οδήγηση να την προκρίνουμε της ε, κατεξουδιώτησης ε, πράξης πρέπει να σας πω πως εδώ θα έπρεπε ε, να τις χρησιμοποιήσουμε και για τις διοξίνες αζότου και τα όρια ανώτα που θα θεσπίσουμε εκεί, αλλά και για κάποιες ε, προτάσεις οι οποίες εάν δεν τοποθετηθούν τα όρια αυτά για το συγκεκριμένο πρόβλημα της διοξίνης αζότου μπορεί να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν πρέπει να καθυστερούμε. Η κατεξοδότηση πράξη είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε να προχωρήσουμε με το γοργό ρυθμό που χρειάζεται και να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο να ασκήσει το δημοκρατικό έλεγχο, να ασκήσει το δικαίωμα βότου, ε, το, ε, με συγχωρείτε, ε, βέτο που έχει, εάν οι προτάσεις δεν μας ικανοποιήσουν. Χρειαζόμαστε μια προθεσμία έτσι ώστε να προχωρήσει και να καταφέρει θέσει προτάσει μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Φώστα. Φώστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ήταν πολύ πλήρης η δουλειά της μέχρι τώρα. Οπωσδήποτε είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει η Επιτροπή Περιβάλλοντος για αυτή την έκθεση. Αυτή είναι η κυρία άποψη το ότι εμείς ε, είμαστε πάρα πολύ θετικοί και θέλουμε περισσότερο την συναπόφαση παρά ε, τη κατεξοδότηση πράξη. Θεωρήσαμε ότι δεν είναι ό,τι πιο σωστό. Θα ήθελα να σα πω για ένα-δύο άλλα πραγματάκια. Ότι δεν συμφωνούμε με κάποιες από τι συμβαστικέ τροπολογίε. Ορισμένε θεωρούμε ότι είναι εντάξει και μερικέ θα τι ψηφίσουμε. Αλλά ακόμη έχουμε πρόβλημα με κάποιες τροπολογίε οι οποίες παραπέμπουν στα νέα όρια εκπομπή για το μονοξίδι του ε, άνθρακα και επίσης ε, άλλες εκπομπές. Γιατί στις χαμηλές θερμοκρασίες δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα τέτοιο πρόβλημα και εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες. Επίσης, για κάποιες άλλες σημαντικές, εκεί που λέει για την υποχρεωτικότητα αυτών των ε, δικτών κατανάλωσης, και όσον αφορά τις ε, αλλαγές ταχύτητος, το σχετικό όργανο. Οπότε, ανάλογα με το τι θα γίνει με τις ε, τροπολογίες, θα δούμε κατά πόσον θα ψηφίσουμε το κείμενο, ανάλογα με το πώς θα αντιμετωπίσουμε πολλά ε, προβλήματα. Και αυτό είναι κρίμα βέβαια, γιατί επί της αρχής συμφωνούμε με το άλλη έκθεση. Να δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα στην έκθεση περιβάλλοντος. Πρόκειται για νομοθέτημα μάλλον περίπλοκο. Ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια. Η κυρία Μάγια, πρόεδρε. Ευχαριστώ την συντάκτη τη νομοδότησης. Είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με, τις, με την προσπάθεια να συγκρατήσουμε ή να μειώσουμε τις εκπομπές ε, που έχουν βλαπτικά ε, σωματίδια. Εμείς δεν συμφωνούμε με τη, γνωμοδότηση, με τη ως προς το μεθάνιο. Γιατί πρέπει να κοιτάμε όχι τα αέρια του θερμοκηπίου, αλλά τα ρηπογόνα σωματίδια. Αυτό είναι το θέμα της γνωμοδότησης. Ξέρω ότι γενικά λένε ότι επειδή επηρεάζει τις κλιματικές ε, συνθήκες ε, και προξενεί κλιματική αλλαγή το μεθάνιο, ε, γενικά περιλαμβάνει τους ρυθμίσεις, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μικροσωματίδια και άρα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί το μεθάνιο ως αέριο του θερμοκηπίου. Άλλο, αν μιλήσουμε για διοξίδιο του άνθρακα, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε μια τελείως διαφορετική, με ένα τελείως διαφορετικό κλάδο της πολιτικής και άρα θα πρέπει να γίνουν μελέτες κτλ. Ε, δεν θα μπορέσουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τη συμβαστική 1. Εκεί θα δείτε ότι και συναδελφοί άλλοι από την άλλη, όχι μόνο εγώ, έχουν διατυπώσει τροπολογίες για να ακολουθήσουμε διαφορετική επιλογή. Επομένως, συμφωνούμε επί της ιδέας ότι πρέπει να περιοριστεί το μεθάνιο, το εκπομπές μεθανίου, αλλά δεν έχει θέση αυτή η ρύθμιση στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Επίσης, ε, στη δεύτερη συμβαστική, αυτή η παράδοξη τάση να ενισχύονται όλο και περισσότερο οι διαδικασίες της κατ' εξουσιοδότηση νομοθέτησης εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι νομίζω υπερβολική. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό και αποκλεισμό του Κοινοβουλίου από τις νομοθετικές διαδικασίες. Μιλούμε για συναπόφαση, συναπόφαση θέλουμε και όχι κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Για τους υποχρεωτικούς μετρητές κατανάλωσης καυσίμων Πάλι υπερβολικό μας φαίνεται. Υπάρχουν ούτως ή άλλως ε, σε μεγάλο βαθμό των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων ε, αλλά και των ε, φορτηγών και άλλωστε είναι και προσφέρον του οδηγού τέτοιου είδους μηχανισμοί. Δεν βλέπω έτσι πρέπει να τα καταστήσουμε υποχρεωτικό. Επίσης για τις εκπομπές πραγματικού χρόνου, νομίζω θα πρέπει να το πούμε, ίσως ο συνάδελφος Φέρθηκε ήδη στις ε, προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει ε, συστήματα προσωμείωσης γνήσιων συνθήκων οδήγησης και πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα ε, τι έχει να μας πει η Επιτροπή όταν θα είναι έτοιμη η δουλειά του και μετά να συζητήσουμε για οποιασδήποτε αξίες. Προδικάζοντας δηλαδή την έκβαση των εργασιών της Επιτροπής. είναι κάτι το οποίο νομίζω ακολουθεί όλη η ομάδα της Άλτα. Ξέρω βεβαίως ότι και εσείς όπως και εμείς θέλετε μια λογική λύση που θα οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και από τα φορτηγά αυτοκίνητα. Ευχαριστώ κύριε Κίλα. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ τεχνική γνωμοδότηση. Δεν θα μπω τώρα στις διάφορες τροπολογίες με λεπτομέρειες. Νομίζω πως έχουμε έναν πιθανό συμβιβασμό και Βεβαίω δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλα τα θέματα όλες οι ομάδες. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό γιατί το θέμα το οποίο συζητάμε δημιουργεί πάρα πολλές ε, προκλήσεις και υπάρχουν και τεχνικά στοιχεία τα οποία είναι αντιφατικά. Για παράδειγμα, ε, οι προσπάθειες που κάνουμε για τη μείωση των εκπομπών θα μπορούσαν να επιτευχθούμε και με διαφορετικές λύσεις, όχι μόνο αυτές που προτείνονται εδώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες λύσεις, οι ηλεκτρονικές συγκοινωνίες, ηλεκτρικές για παράδειγμα, ή διαφορετικό είδος αστικών ε, ε, κέντρων. Επίσης, ε, τι γίνεται με το carpooling, αν μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε πολύ το ίδιο αυτοκίνητο, άλλες προσπάθειες που μπορούν να γίνουν για να προστατεύσουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενναίες. Μην ξεχνάτε πως οι εκπομπές από τα μέσα συγκοινωνίας σκοτώνουν περισσότερους από τα οδικά ατυχήματα. Άρα λοιπόν δεν είναι ε, ίσονο σημασία στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Danke sehr, Well, thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Η μείωση κάθε παράγοντα μόλυνσης, αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Και τα, τα πρότυπα 5 και 6 για την Ευρώπη. Είναι ευκαιρία να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Όμως, όπως σας είπα και την τελευταία φορά, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρει καθόλου μέτρα τα οποία πρόκειται να μειώσουν αυτές τις εκπομπές. Απλώς μειώνει την ευελιξία που έχουν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να συμβούσουμε τις τοπολογίες που αφορούν αυτά τα όργανα μέτρησης κατανάλωσης και της ε, αλλαγής των ταχυτήτων όπως προτείνει η Τώρα, ε, για το GSI, αυτούς δηλαδή, τους, ε, αυτά τα όργανα, αυτούς τους δείκτες, ε, θα μπορούσαν να μειώνουν όμως την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα και με την πρώτη τροπολογία, ε, εκεί που αφορά το μεθάνιο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θα μπορούσε εδώ πέρα να υπάρξει μια αντιστοιχία με την μόλυνση από το διοξίδιο. Και για τα νέα επιβατικά όπως και για τα ελαφρά φορτηγά, να έχουμε κάποιες οριακές τιμές, όπως έχουμε και για το διοξίδιο. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία υπαριθμών 2, δεν θεωρούμε ότι τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν ε, αέριο θα πρέπει να την χάνουν κάποιο μεγαλύτερο περιθωρίο βλαπτικών εκπομπών σε σχέση με τα άλλα οχήματα. Προβλέπω ότι θα υπάρξει αύξηση όσον αφορά ε, τις ε, βλαπτικές εκπομπές από τέτοια οχήματα. Ο Πρόεδρος. είναι έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Όσον αφορά τη, τη λύση για τη μόλυνση, δεν θα τα πράγματα τόσο εύκολα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι ότι τώρα θέλουμε να κάνουμε τη μετάβαση σε καινούργιες μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες κλπ. Παρ' όλα αυτά για όλη αυτή την έκθεση βλέπουμε ότι κάποια στοιχεία είναι αποδεκτά ε, όσον αφορά τη διάταξη για το μεθάνιο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το μεθάνιο όσον αφορά την μέτρηση των εκπομπών. Υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ήδη έχει αναφερθεί. Είναι ε, το θέμα της ε, επιλεγής της διαδικασίας όσον αφορά αυτές τις ε, της πράξης. Δεν νομίζω ότι είναι ότι πιο δόκιμο εδώ για τα μέτρα αυτά για τις εκπομπές το ότι θέλουμε σε κάποια φάση να μην έχει το, το, το κοινοβούλιο την πρωτοβουλία ενεργειών που τη δικαιούται. Άρα ίσως θα πρέπει εδώ να ακολουθηθεί η συνήθιση νομοθετική διαδικασία και γι' αυτό και εμείς κατεβάσαμε κάποιες τροπολογίες ούτως ώστε να ζητήσουμε μια νέα νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη μελέτη των επιπτώσεων. Είναι πολύ γενικό χαρακτήρα αυτή η μελέτη που υπάρχει και συζητήσαμε οι σκιώδεις στην συναντησή μας. Οπότε γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και επομένως αντίστοιχες είναι και τοπολογίες οι οποίες κατεβάσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πίπερ Κούν. Παρακαλώ από ένα λεπτό καθένας πια, γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Κύριος Πίπερ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε πολύ φιλόδοξη στόχοθέτηση για το διοξείδιο του άνθρακα στα, στα οχήματα, στις οδικές μεταφορές και νομίζω ότι μέγα μέρος ε, της ευρωστίας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας οφείλεται σε αυτές τις διατάξεις. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην βαστική υπαριθμόν 1 για, την, για το μεθάνιο. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να αποκλείει το, μεθάνιο, γιατί αν συμπεριληφθεί το μεθάνιο, το οποίο έχει τόσο μικρή, καταρχάς δεν έχει σχέση δηλαδή με τα μικροσωματίδια, και δεύτερον θα ε, καταστεί πάρα πολύ δύσκολος ο υπολογισμός ιονδήποτε τιμών για τον ε, αυτοκίνητο βιομηχανία μας. Θέλω να κοιτάξω λοιπόν ε, το θέμα υπό την σκοπιά του, της αποστολής μας ως Επιτροπής, γιατί εμείς δεν είμαστε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, είμαστε η Επιτροπή Μεταφορών, αν δεν απατώμε, άρα πρέπει να κοιτάμε να διευκολύνουμε τις μεταφορές και, την, ε, και το σχετικό κλάδο. Ε, ας μην ε, ανατρέψουμε ε, διατάξεις ε, που ισχύουν εδώ και χρόνια για την αυτοκινητοβιομηχανία με μια τέτοια διάταξη. Ευχαριστώ κύριο Νίλσον. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε γιατί στις αρχικές μας συζητήσεις μιλήσαμε για επικάλυψη με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το σημαντικότερο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα ανώτατα όρια τα οποία θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα την βιομηχανία και θα ξεκαθαρίσουν το ποιό είναι οι προθέσεις μας. Αλλά θα ήθελα να σας προειδοποιήσω το ότι να συζητάμε εδώ τόσο τεχνικά θέματα και να προσπαθούμε εμεί να νομοθετήσουμε για τεχνικά ζητήματα ενδεχομένως μπορεί να περιορίσει την καινοτομία. Γιατί εάν απλώς επιβάλλουμε αυστηρότερα ανώτατα όρια τότε η καινοτομία θα θριαμβεύσει και είδατε, ε, για παράδειγμα, την, ηλιακή, την ενέργεια τι έχουμε καταφέρει, θεσπίζοντας σοβαρούς κανόνες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπερρυθμίζουμε τα θέματα σε τεχνικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μερικές παρατηρήσεις μόνο, διότι έχει να κάνει βέβαια με τη ρήπανση, το περιβάλλον και την υγεία Η γνωμοδότηση αυτή έχει να κάνει με την εκπομπή δηλαδή ρηπογόνων ε, μικροσωματιδίων. Υπάρχουν και κάποια τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό τους. Εν πάση περιπτώσει εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ανώτατες τιμές. Ε, οξύδια του ε, αζότου που είναι πολύ επιζήμια, επικίνδυνα και φτάνουν μέσω των εκπομπών των οχημάτων να πολλαπλασιάσουν στην ατμοσφαιρική στο ατμοσφαιρικό αέρα γιατί υπάρχει φυσικά άζωτο στο ατμοσφαιρικό αέρα και λόγω των εκπομπών κάνει ενώσεις πολύ επικίνδυνες το μονοξίδιο του άνθρακα βεβαίω, που είναι πολύ επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και έτσι είναι αυτό το θέμα του, της νομοδότησής μας. Από το 2011 και πιο πριν ακόμα, εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, είχαμε προσδιορίσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα σε τα επίπεδα, στα 130 ε, γραμμάρια ανά, χιλιόμετρα, ανά χιλιόμετρο και θα πρέπει αντίστοιχα μέχρι το 2021 να έχουμε φτάσει ε, για κάθε λίτρο βενζίνης ή δίζελ που καίει ένα όχημα ε, στις τιμές αυτές έως το 2021 όπως έλεγα. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε είδους καύσιμο που καίμε μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, αυτό είναι μια γενική αρχή, ε, είναι γνωστό. Ένα λεπτό να σε διακόψω, έχεις περάσει τα δύο λεπτά. Είναι άδικο και πέναντι στους άλλους συναδέλφους. Το λέω λοιπόν, ναι, ναι, ναι, μα είμαι υπομονετικός βεβαίως. Δυστυχώς κυρία Μάισνερ δεν ακούγεται. Ο κύριος Σιμάνσκι λοιπόν, Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, γεια σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να υποβάλει κάποιε συγκεκριμένε παρατηρήσει. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για όλε τι ε, τροπολογίε. Επίση, νομίζουμε ότι είναι προ τη σωστή κατεύθυνση και υπάρχει ένα κοινό παρονομαστή σε σχέση με τη δική μα πρόταση για να έχουμε την μείωση των εκπομπών και επίσης να έχουμε περισσότερη αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Περιμένουμε για να δούμε τι θα προγύψει από τη ψηφοφορία αύριο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αν μπορούσα, θα έκανα δεκτές όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν αυτό. Για το μεθάνιο τώρα, στη συμβαστική υπαριθμόν 1. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε εδώ το εξή, ότι έχουμε πει όχι στις κατεξουσιοδότηση πράξεις και έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πλήρη μελέτη μετά από διαβουλεύσει με τον κλάδο, του κατασκευαστέ κτλ. Δηλαδή, κάθε φορά που η Επιτροπή θα ε, κάνει μια πρόταση την οποία εμείς θεωρούμε ακραία, θα μπορούμε να παραπέμπουμε σε αυτή την απόφαση για τις διαβουλεύσει. Και όπως είπα θα ήθελα να σας ικανοποιήσω όλους σε όλα σας τα μελήματα, τα αιτήματα και τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία όλους και τους ηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, την εισηγήτρια, τους και ηγητές, όσους έλαβαν μέρος. Ψηφοφορία αύριο 10 το πρωί. Επόμενο θέμα. Η παρουσίαση από τον Υπουργό της Λετωνίας για τις μεταφορές, τον κύριο Ανδρέας Μάτης, ο οποίος είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Σας περιμένουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Να ξαναρχίσω λοιπόν, αφού δεν ακογόμουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βρίσκομαι ανάμεσά σα σήμερα για να σα ενημερώσω για το τι καταφέραμε στη διάρκεια τη δική μα Προεδρία. Την περασμένη εβδομάδα οι Υπουργοί Μεταφορών συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο και εκεί συμφώνησαν την γενική προσέγγιση τη πρόταση την ιστοδηγία για τι τεχνικές απαιτήσει για τα σκάφη εσωτερικής ε, ακτοπλοείας. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι και τα κρατημέλη και η Προεδρία έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες για να βελτιώσουν την πρόταση αυτή, για να δούμε γεωγραφικά ποιο πεδίο καλύπτει και για να εντάξουμε ε, και την Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στήριξε στις προσπάθειές μας αυτές. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω πως στις αρχές Ιουνίου η κεντρική ε, Επιτροπή Ναυσιπλοεία σε εννέα κράτη-μέλη συμφώνησε πως είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνώμων και συμφώνησε και τις αρχές επί τις οποίες θα εργάζονται, το οποίο αποτελεί ένα προαπαιτούμενο για να επιτύχουμε μια συμφωνία για να ε, προωθήσουμε την ε, βιομηχανία της Εσωτερική ναυσιπλοεία στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια τελική συμφωνία για την οδηγία αυτή και ελπίζουμε πως ε, έτσι η Ευρώπη θα χρησιμοποιεί όχι μόνο δρόμους αλλά και τις πλωτές οδούς στις προσπάθειες που γίνονται για, τις, την βελτίωση των επιδόσεων των μεταφορών. Τώρα, για τις χερσαίες μεταφορές, η δική μας Προεδρία πρέπει να σας πω ότι προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τους σιδηροδρόμους βασιστήκαμε σε επιτυχίες της Ιταλικής ε, ε, Προεδρίας που κατάφερε να συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσημα εγκρίναμε δύο ε, νομικές πράξεις για τις δάτινες μεταφορές. Έχουμε τα, τα πρόστιμα, τα διασυνοριακά πρόστιμα, όπως επίσης και τις, συγχωρείτε αυτό αφορά τις μεταφορές και τις διαστάσεις των οχημάτων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Τώρα, για την οδική ασφάλεια, να σας πληροφορήσω ότι την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενδιάμεση αναθεώρηση που έγινε για το πλαίσιο της πολιτικής για την οδική ασφάλεια 2010-2020. Καλωσορίζουμε το γεγονός πως η Προεδρία του Λουξεμβούργου επίσης φέτος τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο που θα γίνει τότε σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το θέμα της οδικής ασφάλειας στα πλαίσια της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές. Εάν επιστρέψουμε τώρα στο θέμα των σιδηροδρόμων, τον Ιανουάριο φέτος συνεδριάσαμε για πρώτη φορά για το τέταρτο πακέτο γιατί ήταν ένα από τα κομβικά σημεία κατά τη γνώμη μας για τη δική μας λετωνική προεδρία στο οποίο αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις για τους δύο άξονες αυτού του πακέτου και νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και για τους δύο. Μιλώντας ε, για τον πυλώνα της αγοράς, η Προεδρία, όπως είχε υποσχεθεί, συνέχισε τις προσπάθειες που είχε ξεκινήσει η Ιταλία και προετοίμασε και εξέτασε αρκετά συμβιβαστικά κείμενα και για τα BSO και για τη διαχείριση δικτύων και δεδομένης της πολιτικής ευαισθησίας του θέματος το Συμβούλιο το Μάρτιο παρακάλεσα τους συναδέλφους να με κατευθύνουν. Να μου πούν τι πρέπει να κάνει το Συμβούλιο. Γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Για την πρόταση για τη διαχείριση των δικτύων έχουμε την ανεξαρτησία των διαχειριστών των υποδομών ε, και έχουμε και το θέμα ε, της πρόσβασης ε, στο τροχοφόρο υλικό έγιναν πολλές συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο και νομίζω ότι για τις περισσότερες από τις βρήκαμε λύσεις. από την Προεδρία μας πρέπει να σας πω πως στηριχθήκαμε από διάφορα ε, κινήματα, με συγχωρείτε, από διάφορα κείμενα συμβιβαστικά, ε, τα οποία είχαν ήδη προταθεί από τις αρχές του 2013. Κάνουμε μια αξιολόγηση της έκθεσης προόδου την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών και χάρηκα που άκουσα τους συναδέλφους να λένε πως οι συζητήσεις μέχρι εδώ έχουν καρποφορήσει και θα προσφέρουν σημαντικά στην προσπάθεια που γίνεται να συμφωνήσουν το θέμα αυτό τα κράτη-μέλη, τα οποία, επαναλαμβάνω, συνεχίζουν τις προσπάθειες που κάνουν. Για την επόμενη Προεδρία, ε, τον Υπουργό, τον κύριο Μπόσκ και το Λουξεμβούργο, θα ήθελα να τους εγχαρώ για την επιθυμία που ε, δείχνουν να συνεχίσουν την πολιτική συζήτηση ε, του θέματο αυτού, ξεκινώντα κάποιε συζητήσει όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά και με το Κοινοβούλιο. Τώρα, αν, μιλάμε για, αν μιλήσουμε για το τεχνικό κομμάτι, τον τεχνικό άξονα του πακέτου, εκεί δεν έχουν κλείσει τα θέματα. Πολλέ συζητήσει γίνονται, έχουμε αρκετέ εκκρεμότητε για τι οποίε έχει βρεθεί μια λύση, και πρέπει να σας πω ότι η λύση την οποία προκρίνουμε είναι αυτή που προτιμάει και ο κλάδος. Μια που βρίσκομαι εδώ, εκ μέρους της Προεδρίας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς, τις ομάδες σας για την επικοδομητική συνεργασία. Γιατί είναι θέματα τα οποία και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο είναι περίπλοκα. Την Τετάρτη θα γίνει η έναντι συνάντηση του διαλόγου σε τριμερές επίπεδο και ελπίζουμε πως θα είναι και η τελική. Τα Θέματα που μένουν είναι οι εφαρμοστικέ πράξει, οι κατεξουδότητε πράξει και οι ε, προθεσμίε εφαρμογή που αποτελούν τα τελευταία εμπόδια πριν επιτέλου πετύχουμε το στόχο μα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι εισηγητέ, για το τέταρτο πακέτο, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, σκιώδει εισηγητέ, οι προσπάθειες που κάναμε το περασμένο εξάμεινο μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την αποφασιστική στιγμή. Τα τελευταία βήματα πριν το τέλος θα είναι τα πιο δύσκολα, το γνωρίζω. Παράλληλα είναι στα χέρια μας να πετύχουμε μια συμφωνία. Μην ξεχνάτε ποιο είναι ο ουσιαστικό στόχο του τεχνικού σκέλου αυτού του πακέτου, δηλαδή να στηρίξουμε τη βιομηχανία μα στο θέμα αυτό. Δεδομένη τη κατάσταση στη διεθνή αγορά, είναι ξεκάθαρο και πασιφανέ θα έλεγα Πώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση όπω αυτή εξελίσσεται και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να προσφέρουν μια ουσιαστική στήριξη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των σιδηροδρόμων. Πιστεύω, συνάδελφοι, πως μπορούμε να λύσουμε το θέμα που μένει πια σε κρεμότητα στον τριμερή διάλογο που θα κάνουμε τούτη εδώ την εβδομάδα. Μετά έχουμε και κάποια θέματα ε, αεροναυσιπλοείας. Εκεί ανεξέθετα από τις δυσκολίες συνέχισε τις συζητήσεις η Προεδρία για τα όσα είχαν ξεκινήσει η Ελληνική και μετά η πολυφανική προεδρία για τα δικαιώματα των επιβατών. Και εκεί να σας πω πως κάναμε κάθε προσπάθεια για να βρούμε ένα συμβιβασμό για τα θέματα που είναι σε κρεμότητα και μάλιστα καταφέρουμε αρκετά. Όμως παρόλου τους συμβιβασμούς που προτάθηκαν από την Προεδρία, το θέμα δηλαδή του ορίου αποζημίωσης σε περίπτωση που έχει χάσει κανείς την επόμενη πτήση και το θέμα του Γιβραλτάρ παραμένουν ανοιχτά. Γιατί βέβαια και το Γιβραλτάρ επηρεάζει πάρα πολύ τα δικαιώματα επιβατών και ελπίζω πως θα το αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Και ελπίζω πως θα μπορέσει να συμφωνήσει το Συμβούλιο ένα συμβιβασμό που θα καλύπτει αφενός τα δικαιώματα των επιβατών, αφετέρου τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Για το Γιβραλτάρ τώρα, τι να πω. Περιορισμένη η, πρόεδρος που έχει, η πρόοδος που έχει γίνει. Και είναι πολλές οι για τον κλάδο εδώ. Αυτό που θα θέλαμε εμείς να προσφέρουμε στις συζητήσεις που γίνονται για τις στρατηγικές προτεραιότητες του κλάδου, τις οποίες στηρίζει ο κλάδος. Να σας πω πως 13 του μηνός έγινε μια προσπάθεια να γευματίσουμε εμείς εδώ με εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου και με του κλάδου και να πούμε πως έχουμε τρεις προτεραιότητες. Καταρχήν, η εξωτερική και εσωτερική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπλοείας. Δεύτερον, ανάπτυξη και απασχόληση. Και τρίτον, διαλειτουργικότητα για τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα στην Ευρώπη. Για το πρώτο θέμα, οι Υπουργοί μίλησαν για το διοικητικό άχθος, όπως επίσης και το ποια μπορεί να είναι η κρατική ενίσχυση που προσφέρεται στα αεροδρόμια. Γιατί θα πρέπει να έχουμε καταρχήν το απαραίτητο δυναμικό σε επίπεδο υποδομών, θα πρέπει να κάνουμε πιο ανταγωνιστικούς τους Ευρωπαίους αερομεταφορείς και αυτό σε σύγκριση με τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών και βεβαίως θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις που γίνονται τις προσπάθειες για ανάπτυξη και απασχόληση. Τεχνολογία, καινοτομία, υποδομές, τα γνωστά θέματα που μας απασχολούν. Τώρα, εσωτερική διαλειτουργικότητα, κρίσιμο σημείο για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Όχι μόνο να ενισχύσουμε τα μεγάλα αεροδρόμια κόμβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να ενισχύσουμε και τη διαλειτουργικότητα ε, στις διάφορες συνδέσεις που έχουμε με τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ευρώπης. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πως είναι το έτος της αεροπλοείας και αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν ένα νέο πακέτο για να καταθέσουν και ελπίζω πως θα λάβουν υπόψη τα στρατηγικά αυτά θέματα τα οποία έχουν θέσει τα κράτη-μέλη. Επειδή όλο ένα αυξάνονται ε, οι δυνατότητες που έχουν τα ντρόουν και τα, τηλεκατευθυνόμενα ε, αεροπλάνα, οργανώσαμε μία εκδήλωση για αυτά τα ντρόουν ή τα τηλεκατευθυνόμενα στη Ρήγα και εκεί συζητήσαμε τις προκλήσεις που έχουμε σε αυτό τον κλάδο που αναπτύσσεται όλο ένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε την ανακοίνωση λοιπόν τη δήλωση της ε, Ρήγας που εγκρίθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής μια σημαντική κατάθεση και συνεισφορά σε κανονισμό που θα φαντάζομαι προετοιμάσουμε στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και στα θέματα της εξωτερικής ε, πολιτικής αεροπλοείας, δηλαδή συμφωνίες ασφάλειας ε, με την ΙΠΑ, με την Βραζιλία, με την Κροατία. Μία ακόμα προτεραιότητα είναι το Engage Europe. Τέλη Απριλίου στη Ρήγα έγινε μια συνάντηση υπουργικό επίπεδο όπου εγκρίθηκε και πάλι μια δήλωση της Ρήγας όπου αναφέρεται στο πώς θα με τα κράτη-μέλη στις αερομεταφορές να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα ε, συστήματα χερσαίων μεταφορών για ε, λειτουργικές ε, λύσεις που θα συνδέσουν την Ασία με την Ευρώπη. Να διευρύνουμε τα δίκτυα μεταφορών, μια και αυξάνεται συνέχεια το εμπόριο της Ευρώπης με την Ασία και για τους χερσαίους διαδρόμους για την ε, ε για τα υπηρετικά σύνορα Ευρώπης-Ασίας να σας πω πως έχουμε εδώ κάποιους σιδηροδρόμους οι οποίοι διασχίζουν ολόκληρη την περιοχή αυτή οι οποίοι θα πρέπει να ισχυθούν. Έχουμε τα δίκτυα TNT και έχουμε επίσης και τους διαδρόμους για τα θέματα αυτά το Μάρτιο ε, συζητήσανε οι Υπουργοί τα θέματα αυτά γιατί οι επενδύσεις για παράδειγμα στην στρατηγική για την αιτής ανάπτυξη ε, είναι σημαντικό θέμα και συζητήσαμε τι γίνεται με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπως επίσης και με τη στρατηγική για το 2020. Βασική... Βασικός άξονας είναι το πώς μπορεί να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πώς μπορούμε να προσφέρουμε θέσεις απασχόλησης, και βρήκαμε μια ευκαιρία έτσι ώστε οι Υπουργοί Μεταφορών να συζητήσουν ε, την ευρύτερη διάσταση αυτών των ε, προβλημάτων. Τώρα, το επενδυτικό σχέδιο Juncker. Εδώ θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε έτσι ώστε ο χώρος των μεταφορών να είναι πολύ ορατός στα πλαίσια αυτού του πακέτου. Που θα αρχίσει ήδη να μοιράζει κονδύλια από το φθινόπωρο. Οι πιο λεπτομερεί συζητήσει για τα δίκτυα TNT έχει να κάνει με τις ε, επενδύσεις, με εναλλακτικά σχέδια και την επόμενη εβδομάδα στη Ρήγα έχουμε οργανώσει αυτές τις ημερίδες TNT ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε τα σχετικά θέματα. Θα κλείσω ευχαριστώντας και πάλι ε, και εσά κύριε Κράμερ αλλά και όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής για την τόσο επικοδομητική συνεργασία και ελπίζω πως αυτή την εβδομάδα εσείς και εμείς στη Λετωνική Προεδρία θα κάνουμε και αυτό το τελευταίο βήμα που θα μας οδηγήσει στο αίσιο τέλος. Και εύχομαι βέβαια και κάθε επιτυχία στο Λουξεμβούργο που έπεται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ. Πολύ ευχαριστώ. Ανταποδίδω και εγώ τι ευχαριστίε εκ μέρου όλων των εμπλεκομένων. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά η Λετωνική Προεδρία σε σχέση με τον τριμερή διάλογο για, τον, ε, για το πακέτο για του σιδηροδρόμου. Ήταν για μα μεγάλη πηγή ικανοποίηση, στάση τη δηλαδή. Έχουμε όμω κάποια άλλα θέματα που ελπίζω να προχωρήσουμε έτσι ώστε να είμαστε όλοι ικανομένοι. Και πάντα το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικό από ότι ο χρόνος Δίνω το λόγο στους συντονιστές, ο κύριος Φανταρκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη έκθεση όσον αφορά την αξιολόγηση της Λετωνικής Προεδρίας είναι θετική. Παρακαλώ να τα πρακτικά Βεβαίως και δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ούτε ε, ακόμα βέβαια ολοκληρώθηκε η Προεδρία, αλλά έχουν κάθε λόγο να δέχονται συγχαρητήρια οι προεδρεύοντες κοινότητες. Επίσης βοήθησαν τα επιτεύγματα της Ιταλικής Προεδρίας, αλλά δεν είχαν γίνει και τόσα πολλά. Αλλά σίγουρα οι ρίζε της επιτυχίας έγκυται σε εκείνη την Προεδρία. Και ήταν ε, πάρα πολύ θετικό το ότι άρχισε ε, την εισήγησή του ο κύριος Υπουργό με τι ιστορικές πλωτέ οδού, γιατί χρειάζεται εκεί ε, προσαρμογή τη ε, νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνικές διατάξεις για αυτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και όσον αφορά τον Ρήνο, αλλά όσον αφορά και τον Δούναβιου είναι πολύ σημαντικά αυτά. Τώρα προς το τέλος. leveren. En bij de komende raadspresident. Μα ενδιαφέρει βεβαίω και το πακέτο Juncker. Αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς θα υπάρξουν επενδύσεις στρατηγικές και στις μεταφορές. Την Τετάρτη θα υπάρξουν κάποιοι σκόπελοι στο Συμβούλιο, ελπίζουμε ότι όσον αφορά τις ε, τεχνικές πράξεις και τις μεταβατικές περιόδους, ότι θα γίνει ό,τι πρέπει. Ε, τότε θα έχετε ακόμη περισσότερα τρόπια σαν Προεδρία με το παιδί και αυτό. Το θέμα είναι γιατί δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα κάποια κοινή προσέγγιση. Τι γίνεται με την πολιτική πτυχή των πραγμάτων οι ψήφοι στου διαδρόμου λένε ότι έχετε σημαίνει πρώτα τον Ιούνιο δεν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο σα και θα πρέπει να περιμένουμε οι Λουξεμβούργοι να ολοκληρώσουν το έργο σα Τώρα, όσον αφορά την αεροπλοεία, είναι μάλλον τραγικό ότι κατά το εξάμεινο της Προεδρίας σας δεν καταφέραμε και τίποτα. Υπήρξε και αυτό το σοβαρό πρόβλημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας. Αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι ε, μια αφετηρία δράσης για την επόμενη Προεδρία. Οπότε και θα καταστεί δυνατόν να συνεχιστεί το έργο σας. Πάντως σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Και για ακόμα μια φορά είδαμε ότι οι μικρές χώρες καταφέρουν περισσότερο από ότι οι μεγάλες στην Προεδρία. Ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ Ισμαήλ Ερτού. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Υπουργέ, ήθελα προσωπικά αλλά και εκ μέρους της ομάδας μας σας ευχαριστώ για το τελευταίο αυτό εξάμεινο της συνεργασίας ε, στο πεδίο των εργασιών μας. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι η δουλειά σας έγινε με τρόπο ψύχρεμο, αποτελεσματικό και όπου υπήρχε η δυνατότητα διαπιστώνω ότι επιλέξατε διατυπώσεις τέτοιες οι οποίες ήταν αποδεκτές για κάθε πλευρά. Βεβαίως υπάρχουν ακαθόδη ζητήματα, κάποια ήδη αναφέρθηκαν και εσείς στην ομιλία σας αναφερθήκατε για το τέταρτο ε, πακέτο σιδηροδρόμων. Ήταν ε, βεβαίω αναμενόμενο, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, σημαντικό για τα κράτη-μέλη, με διαφορετικές προτεραιότητες για το κάθε κράτος μέλος. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο δηλαδή. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε στον τομέα του τέταρτου αυτού σιδηροδρομικού πακέτου και κυρίως ως προς τα τεχνικά πακέτα, τα τεχνικά θέματα, όπου πιστεύω ότι έχει γίνει πρόοδος όντως. Και νομίζω ότι μετά την Προεδρία σας, όταν αναλάβει προ... την Προεδρία του Λουξεμβούργο, τέταρτη κατά σειρά εναλλασσόμενη Προεδρία που θα ασχοληθεί με το τέταρτο αυτό πακέτο σιδηροδρόμων, ελπίζω να προχωρήσουμε περισσότερο. Πάντως εσείς έχετε επιτύχει πολλά. Αναφερθήκατε στα τεχνολογικά ζητήματα. Και την, ε, τα τεχνικά μάλλον ζητήματα, νομοτεχνικά ζητήματα και ως προς τα implementing acts, πράξεις εφαρμογής αλλά και ως προς την ε, περίοδο προσαρμογής, η μεταβατική περίοδο υπάρχουν ζητήματα στα οποία ε, χρειάζονται πιο σαφείς διατυπώσεις για ορισμένα κράτη-μέλη τουλάχιστον και γι' αυτό περιμένω την επόμενη εβδομάδα να εξευρεθεί μια διατύπωση η οποία θα είναι δυνατό να γίνει δεκτή σε επίπεδο Συμβουλίου. Επίσης, Πιστεύω ότι στα πολιτικά ζητήματα η Λουξεμβουριανή Προεδρία πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά, όπως άλλωστε έχει προεξαγγείλει. Θα την υποστηρίξουμε, θα την υποστηρίξετε και εσείς φαντάζομαι, ώστε όταν ολοκληρωθούν αυτά τα τεχνικά ζητήματα να μπορούμε να προχωρήσουμε, δίνοντας όλη μας την προσοχή πλέον στα πολιτικά εκκρεμή ζητήματα στο τέταρτο πακέτο των σιδηροδρόμων. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σημειώσω πως θεωρώ πως δεν είναι ούτε φιωές, ούτε πολιτικά δίκαιο. Τα τεχνικά αυτά ζητήματα που έχουν κλείσει, που θα κλείσουν την επόμενη εβδομάδα, να μην τεθούν σε εφαρμογή, να μην προχωρήσουν δηλαδή. Και θα το πω, να τεθούν σε ομοιρία τα τεχνικά αυτά ζητήματα μέχρι ότου εξευρεθεί η πολιτική λύση στα υπόλοιπα ζητήματα που αναφέρατε και εσείς, το governance, δηλαδή διακυβέρνηση και την, ε, το άνοιγμα των αγορών στις ε, μεταφορές επιβατών. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει επιδείξει μεγάλη υπομονή τους, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων προεδριών. Εγώ προσωπικώς θέλω να σημειώσω ότι καταληκτική προθεσμία για την επεξεργασία των, τεχνο, ζητημάτων θα πρέπει να είναι η 8η Οκτωβρίου με το Σύμβουλο των Υπουργών. Αυτή είναι η κατά βάση πεποίθησή μου, αν και θα επιθυμούσα πολύ ταχύτερη διαθέτηση. Αν όμως ε, δεν θέλουμε να ε, υπάρξει εμπλοκή σε σχέση με τα πολιτικά ζητήματα, καταληκτική προθεσμία πρέπει να, είναι η 8η Οκτωβρίου. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Ύστερα από τέσσερι προεδρίε εναλλασσόμενε, πρέπει πια να είμαστε σε θέση να δώσουμε σαφή μηνύματα στον κλάδο για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει σε νομοτεχνικό επίπεδο και που πρέπει να μπουν πια στο φάκελο. Κάτι ακόμη για το FC τώρα, για το σχέδιο Juncker. Οι δύο συγγητές μας, η κυρία Γιάλα Σέντερ και ο κύριος Ρικέ, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά υπό τις συνθήκες που γνωρίζουμε όλοι εδώ και ένα εξάμεινο. Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει αρκετά γρήγορα για να διατυπώσει μια λύση, μια πρόταση λύσης με για την υλοποίηση του σχεδίου Juncker όπως ονομάζεται, μια σαφή δηλαδή ε, διευκρίνηση. Εγώ προσωπικώ και ω ομάδα δεν είμαστε υπέρ του σχεδίου Juncker με αυτού του όρου. Για να μην με παρεξηγήσετε, θα σα πω ότι θα έλω ένα σχέδιο Juncker το οποίο να έχει σημαντική προσθέμενη αξία. Και επίση θέλω να τυπώσω την επίκριση ε, ω προ το ότι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προχωρήσει χέρι με χέρι και δεν έχουν απαραίτητα παρουσιάσει, τουλάχιστον ω προ τι δικέ μα ε, αξιολογήσει, τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Και όταν ε, έχουμε να κάνουμε με τους προϋπολογισμούς ή τα κονδύλια τα σχετικά με το μέλλον όπως ονομάζονται, τα κονδύλια του μέλλοντος, μεταφορές, τεχνολογία, ε, ευρυζωνικότητα, όλα αυτά για να χρηματοδοτηθούν παίρνουν λεφτά από το Connecting Europe, χωρίς βέβαια αυτό να διευκολύνει την κατάσταση. Ο Ορίζον 2020 έχει χαμηλότερα ποσά από τα 70 δις αν δεν απατώμε που είναι ο μεγάλος προπολογισμό το μεγάλο πακέτο για την επόμενη επταετία. Δεν έχει κανένα νόημα να βάζουμε το ένα κονδύλιο σε ανταγωνιστική σχέση με το άλλο. Δεν είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση και πρέπει να φροντίσουμε τα κριτήρια με βάση τα οποία διοχερτεύονται τα ποσά για το Connecting Europe ε, τα τελευταία δύο χρόνια, τα ποιοτικά αυτά κριτήρια να παραμένουν ενισχύ και με το σχέδιο Juncker των αρχιερών ελληνοποίηση. Για δε τη Λουξεμβουριανή Προεδρία εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά του στην στο επόμενο εξάμεινο. Η ομάδα μου θα είναι πάντοτε σε επαγρύπνηση επικοδομητική και θετική. Ευχαριστώ πολύ. Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τη Λετωνική Προεδρία. Δεν θα σχολιάσω με μεγάλες λεπτομέρειες το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ τον ε, κύριο Σίλερ που το τελευταίο διάστημα είναι στις επάλξεις προσπαθώντας να βοηθήσει τους ε, συναδέλφους να προωθήσει το θέμα. Ξέρω πως έχετε πετύχει κάποια πρόοδο, αλλά βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολο και υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος μπροστά μας. Για τις εσωτερικέ πλωτούς οδούς θα συνταχθώ και εγώ με τους συναδέλφους από κάποια κράτη που έχουν τέτοιες πλωτούς οδούς και που δεν χρησιμοποιούνται παρκώς τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι κάθε είδος συγκοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ό,τι υπάρχει να χρησιμοποιείται και όταν υπάρχουν υποδομές καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται. Κυρίως όταν προσπαθούμε να μεταφέρουμε κάποια εμπορεύματα τα οποία δεν χρειάζεται απαραίτητα να κυκλοφορούν με ε, σιδηροδρόμους ή με φορτηγά. Για τη διασυνοριακή ε, ενημέρωση κανείς δεν θέλει να έρχονται στη χώρα μας άνθρωποι και να ε, παρεβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μετά να λένε ότι αφού φεύγω από τη χώρα ξέφυγα και δεν χρειάζεται ε, να κάνω τίποτα. Ξέρετε πως όταν αλλάζει κανείς νομικό σύστημα πολλές φορές δυσκολεύεται με την επιβολή των προστήμων οπότε η προσπάθεια είναι πολύ καλή. Τώρα για το πακέτο για την αεροναυσιπλοεία ναι, μιλήσατε για την ανακοίνωση, τη δήλωση με συγχωρείτε της ε, Ρήγας και εγώ ε, μιλώ για την πολιτική χρήση αυτών των μη επανδρομένων τηλεκατευθυνωμένων ντρόν και τα λοιπά και εμείς και η ΙΠΑ αναγνωρίσαμε πως αυτή είναι μια τεράστια αγορά που διευρύνεται συνέχεια και αποτελεί και το επόμενο βήμα στο μέλλον της ε, αεροπλοείας. Χαίρομαι λοιπόν που το έχω αναλάβει, είναι μεγάλη πρόκληση, δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν και συνεργάζομαι στενά με τους συναδέλφους για να βρούμε κάτι το οποίο θα είναι πετυχημένο, αλλά αυτό είναι για αργότερα φέτος. Είναι κρίμα, γιατί είχαμε κάποια θέματα τα οποία καθυστέρησαν, είναι κρίμα για το γεγονός πως ο ενιαίος ε, ευρωπαϊκός ουρανός, εθέρας, ε, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, το Single European Sky δεν έχει εμφανιστεί στη συζήτηση. Γιατί εσείς μεν αναφερθήκατε για στο Γεβραλτάρ και εδώ πρέπει να σας επαναλάβω πως δεν έχουμε πρόβλημα με το Γιβραλτάρ. Είναι ε, κράτος υπό την κυριαρχία της Βρετανίας, με αρχηγό κράτος την Βασίλισσα, άλλα κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με το Γιβραλτάρ. Άρα όταν ξεκινήσαμε με τα δικαιώματα των επιβατών στον ενιαίο ευρωπαϊκό εθέρα είχαμε τότε την κυρία Λογιόλα Ντεπαλάσιο, επίτροπο από την Ισπανία. Εγώ ήμουν εδώ, σε τούτη εδώ την επιτροπή στο Κοινοβούλιο και κανεί τότε δεν, είπε, δεν είπε ότι υπάρχει θέμα με το Γιβραλτάρ. Και πέρασαν 10 χρόνια και έχουμε αυτή την γελία κατάσταση η οποία θα πρέπει να επιληθεί. Και νομίζω πω κάποιοι θα πρέπει, πραγματικά κάποιοι, ε, να ανοίξουν τα μάτια του και να δουν ε, αυτή η συμπεριφορά του τι ε, έχει προκαλέσει. Και ξέρετε πως αυτό συμβαίνει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εμείς θέλουμε ο ενιαίος αυτός ευρωπαϊκός εθέρας να προχωρήσει και να δούμε και το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών. Οπότε θα ήθελα να κλείσω λέγοντα ευχαριστώ πολύ την Λετωνική Προεδρία εκ μέρου δική μα πολιτική ομάδα για όσα καταφέρατε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι τα αφήσατε στην καλύτερη δυνατόν κατάσταση δεδομένων των πιέσεων που αντιμετωπίσατε. Ε, θέλουμε λοιπόν και του επόμενου μήνε να διατηρήσουμε την επαφή που είχαμε. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Μάσινερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των φιλελευθέρων θέλω να σα ευχαριστώ και εγώ για όσα κάνατε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία πρώτη σας Προεδρία. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να κάνει σε πρώτη Προεδρία ένα νέο κράτος μέλος. Καταφέρατε πολλά πράγματα, είχατε δύσκολη περίοδο να διατρέξετε. Θα αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα μόνο, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω τα πάντα, αλλά θα επαναλάβω από το λόγια του κυρίου Φαντανκάμπ τις, ε, τους επένους για την αυσιπλοεία. Έχετε καταφέρει σημαντικά πράγματα. Κάποια κράτη, όπως και η Γερμανία εξάλλου, έχουν ε, πλωτές, εσωτερικές πλωτές αλλά, ε, οδούς, αλλά όχι και ως εκ τούτου να με ενδιαφέρονται τόσο πολύ, στους ε, σιδηροδρόμους. Προχωρήσατε ένα φάκελο με ζητήματα δύσκολα. Υπήρξαν βέβαια περιστάσει όπου το κοινοβούλιο δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο και θεωρώ ότι δεν φταίγατε εσεί, δεν χρειάζεται να καταγγείλω τώρα το κράτη-μέλη, το κράτο μέλο που είχε προξενήσει τι δυσκολίε. Πάντω η Λετωνία δεν, έφταιγε. Ε, εσείς κάνατε ότι προούσατε για να διαπραγματευτείτε με τον τριμερή διάλογο, μέσα στον οποίο ασφαλώ πρέπει να εκφραστεί η θέση της πλειονοψηφία. Ε, δεν ολοκληρώθηκαν βέβαια τα θέματα για τι εναέριε ε, μεταφορές. Υπάρχει δυσκολία σχέση με το Γιβραλτάρ. Όλοι θέλουμε τους ενιαίους ε, ευρωπαϊκούς εθέρες και δεν πρέπει το Γιβραλτάρ να καταστεί η πέτρα του σκανδάλου, το ΣΥΠΗΝ στην υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι δυνατόν είτε με το Ηνωμένο Βασίλειο είτε με την Ισπανία να βρεθεί μια λύση ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτω του ποιο έχει τα δικαιώματα εθνική κυριαρχία ή τα κυριαρχικά δικαιώματα καλύτερα πάνω στο βράχο του Γιβραλτάρ. Ε, όλα αυτά νομίζω τα θέματα των μεταφορών μπορούν ανεξαρτήτως να επιληθούν. Για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη drones, ε, συγχαρητήρια, αυτό μόνο μπορώ να πω. Κάνατε καταπληκτική πρόοδο στη Ρήγα, το είδαμε αυτό, σε πολλούς τομείς. Ε, νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις. Για τα TNT, SEF και το EFSI βέβαια, το σχέδιο Juncker, ε, είπατε ότι θα πρέπει να λάβουν ε, πρωταρχική θέση μεταφορές στο σχέδιο Juncker και βεβαίως αναμενόμενο μια και στο Υπουργό των Μεταφορών. Από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί το TNT, ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών δηλαδή και το ε, Ταμείο έχουν πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να ανατραπούν από το σχέδιο Juncker. Έτσι λοιπόν, εμείς βεβαίως υποστηρίζουμε ιδιαιτέρως τις αποφάσεις αυτές που έχουν ε, διαμορφωθεί από ε, τρία θεσμικά όργανα από κοινού. Με το σχέδιο Juncker ε, ξέρουμε ότι μπορεί να εισρεύσει περισσότερο χρήμα από ιδιωτικέ πηγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στόχευση για τα έργα και τις υποδομές που θέλουμε να αναπτύξουμε. Οι μεταφορές έχουν να ωφεληθούν τα μάλα, εάν μπουν σε κύρια γραμμή προτεραιότητας. Εσείς ως υπουργό Μεταφορών δεν ξέρω πώς μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να προσελκύσετε και τους ιδιώτες ε, επενδυτές που χρειάζονται ώστε να αντιληφθούν και αυτοί ότι ε, μπορεί να τους συμφέρει να κάνουν επενδύσεις και στον χώρο των μεταφορών, ταϊρώντας βέβαια τους κανόνες που έχουμε ορίσει. η Νέσα ε, ο Ντομινίκ και η Νέσα έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτό και θα ήταν καλό πιστεύω να μπορέσουμε να διαγνώσουμε αρκετή πρόοδο όταν έρθει η ώρα για την υλοποίηση του σχεδίου Juncker. Ευχαριστώ κυρία Κίλιονεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Λετωνία. Η προεδρία της ήταν πολύ πετυχημένη είχαν τη θέληση να προωθήσουν τα θέματα. Δυστυχώς σε πολλά μέτωπα υπήρχαν ε, κάποιοι οι οποίοι φρέναραν την Προεδρία, αλλά δεν φταίνε η Λετωνοί γι' αυτό. Το τέταρτο πακέτο για τους διαδρόμους ήταν ε, μια διαδρομή που την παρακολούθησα αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι σε αυτό το μέτωπο χάσαμε το τρένο της πρόοδου. Δεν είμαστε στο σημείο που θα έπρεπε να βρεθούμε. μείναμε πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που κατάλαβε το πόσο κανείς θα πρέπει να προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη δεν το κατάλαβε αυτό. Χάσαμε τον χρόνο μας σε διαπραγματεύσεις. Δεν ανταποκριθήκαμε στις ε, προκλήσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε εδώ στην Ευρώπη ότι εμεί οι ίδιοι είμαστε το κύριο εμπόδιο να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Μόλι αυτό αλλάξει, τότε θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία. Με το ενιαίο ουρανό, ήταν ένα άλλο θέμα, το Γιβραλτάρ, και αυτό κράτησε πολλά χρόνια. Οπότε Νομίζω ότι τελικά να έχουμε μια ενιαία ρύθμιση για την ε, αεροπλοεία. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Θα βοηθήσει και την ίδια την αεροπλοεία για αυτό το μέλλον τη στην Ευρώπη. Έχουμε ένα όνειρο. Να έχουμε ενοποίηση των μεταφορών κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα. Άρα ας συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτό τον κοινό στόχο και πάλι να ευχαριστήσουμε την ε, Λετωνική Προεδρία για το έργο της. Προσπάθησαν για τους κοινούς στόχους. Πολύ θετικό αυτό για όλη την Ευρώπη. Και ξέρω αυτοί που ήταν αντιμέτωποι τον πρώτο τι εξελίξει, τώρα τελικά θα συνεργαστούν για το κοινό καλό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Καλή Μαντελή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ και οι οικολόγοι να σας ευχαριστήσουν για ό,τι επιτελέσατε. Ίσως αυτό σας φανεί κάτι το ασυνήθιστο, αλλά σας ερωτώ. Από πλευράς δυσκολιών, τι απολύγισμο θα μπορούσατε να κάνετε όσον αφορά τα διακυβέρματα. Γιατί ε, σήμερα που ε, ολοκληρώνεται η Προεδρία, για πέστε μας, τι συνεργασία θα υπάρξει με την ε, Λουξεμβουργιανή Προεδρία, γιατί μας είπατε ότι έχετε ε, όσον αφορά το χρωτοφυλακείο σας σημαντικά διακυβέρματα και οι συναδελφοί ήδη είπαν πόσο σημαντικό είναι το τέταρτο πακέτο για τους δρόμους ε, και ιδίως από πολιτικής πλευράς. Όπω είπαν λοιπόν οι προελίσσαντε, έχουμε και το σχέδιο Γιούγκερ στις επενδύσει και θα πρέπει τον κύριο Ρικέ και την κυρία Γιάννη Σέντερ να τους ευχαριστήσουμε αλλά για πέστε μα, εσεί τι όραμα έχετε σε σχέση με τα όσα έχετε διαπραγματευτεί για τις ε, ε, μεταφορές Θεωρείτε θετικό ότι σε αυτή τη δέσμη μέτρων υπάρχει κάτι για την ε, βιώσιμη κινητικότητα, τι γίνεται με τους ε, στόχους ε, του να έχουμε συνδρόμους πιο βιώσιμους, ε, είπαμε για τις ιστορικές πλωτές οδούς κλπ. Και μας μίλησατε για την οδική ασφάλεια. Δεν ξέρω, θα, θα τους εκνευρίσω όλους σήμερα, αλλά για πέστε μας εσείς, δεν νιώσατε συγκλονισμένος όταν ακούσατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την εγκατάλειψη των σοβαρά τραυματιμένων στο δρόμο εν ώψη των ρυθμίσεων για το 2020. εσεί ως Προεδρία τι είπατε. Έχουμε αυτό το στόχο, αλλά πώς θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα σχετικά με τι προτάσει της Επιτροπής. Άρα εσείς για πετε μας, τι προσπάθειε θα έπρεπε να καταβάλλετε σε συνεργασία και με την Λουξεμβουργιανή Προεδρία. κυρίω σε τέτοια σημαντικά ζητήματα όπως το Γιβραλτάρ αλλά και γενικότερα τις μεταφορές τις εναέριες μεταφορές για δικαιώματα των ε, ε επιβατών, τα σλότ, τα αεροδρόμια κλπ. Και κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε 6 μήνες έχουμε αυτήν την ε, διάσκεψη για το περιβάλλον και εκεί θα εξεταστεί το θέμα των μεταφορών σε σχέση με το κλίμα. εσείς στη συνεργασία με την επόμενη Προεδρία τι συνεργασία έχετε κάνει. Και κατακλείδη δεν νιώθετε απογοητευμένος για το ότι όσον αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ δεν προχωρήσαμε και τόσο. Ήταν προτεραιότητά μας κατά την Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε πώς θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε ε, και να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Να σχολιάσω το θέμα της οδικής ασφάλειας. Είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ, παρόλο που είναι σημαντικό κοινωνικό dumping, για παράδειγμα, το τι συμβαίνει σε καθημερινό επίπεδο με οδηγούς οι οποίοι δεν αμείβονται αρκετά και οδηγούς οι οποίοι χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες ή άδειε οδήγηση, Τι γίνεται με όλα αυτά, πώς αποφεύγουν ας πούμε, τους ελέγχους. Πρέπει τα θέματα αυτά να τα εντάξουμε στη συζήτηση που γίνεται για την οδική ασφάλεια, γιατί τελικά εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Oui, ce sera très rapide. Γρήγορα να πω πως όπως είπε και ο, συνάδελφος ευχαριστώ την ε, Προεδρία για το τεχνικό κομμάτι στο πακέτο των σιδηροδρόμων. Πολλές συναντήσει. συναντήσεις και ελπίζω πως η συνάντηση θα γίνει σε δύο, μέρος, σε δύο μέρες θα είναι η τελική. Εμείς θα το προσπαθήσουμε. Να επαναλάβω λοιπόν τι ευχαριστήσει τα όσα κάνατε που δεν ήταν απλά στη συζητήση με όλα τα κράτη-μέλη για να καταλήξει σε προτάσεις οι οποίες επιτρέπουν να έχουμε ένα συμβιβασμό αποδεκτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και ελπίζω το αργότερο τον Οκτώβριο να έχουμε κλείσει τουλάχιστον με τον τεχνικό πυλώνα του πακέτου. Ο κύριος Τελέτσκα. Νομίζω πως είχατε δύσκολους φακέλους κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας σας και τους αντιμετωπίσατε με έναν τρόπο που πραγματικά μας ικανοποιεί. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Τα είπαν και οι συνάδελφοι. Να τονίσω κάτι στο οποίο και άλλοι στάθηκαν. Χρειάζομαι να επαναλάβω τα όσα α, ακούστηκαν για το πακέτο Ιούγκερ έχουμε μία υποεκτίμηση του τι θα συμβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες και είναι μάλλον αρνητικό μήνυμα προς τις αγορές. Δηλαδή, έχουμε αποσπάσει τα οικονομικά μέσα από έργα τα οποία δεν θα έχουν αποδόσεις, ε, και το κάνουμε αυτό για να αυξήσουμε την ιδιωτική χρηματοδότηση. Μα νομίζω ότι ο τρόπος που έχουμε επιλέξει είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και υποσκάπτει και τους πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται τα έργα TNT. Εν πάση περιπτώσει, χύθηκε καρδάρα με το γάλα, τώρα τι να πω. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στις κρατικές ενισχύσεις για τις τρίτες χώρες και τους ε, αερομεταφορείς της χώρες αυτές. Μια σκέψη λοιπόν, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για το φάκελο αυτό για την επόμενη Προεδρία. Και τέλος, έχω απόλυτη κατανόηση για το ότι προφανώς δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να μπούμε σε λεπτομέρειες για τα θέματα TNT. θα εκτιμούσα ιδιαίτερα το να μας δίνετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Είσαστε και υπουργό Κοινωνιών, δεν είσαστε μόνο εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και τι θα κάνετε για να ε, ολοκληρώσετε την ε, απορρόφηση των βαλτικών χωρών στο θέμα αυτό από την υπόλοιπη εσωτερική αγορά και πείτε μου ακριβώς τι έχετε στα σκαριά για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να συμφωνήσω με όλου του αδέλφους οι οποίοι ευχαρίστησαν την Λετωνική Προεδρία για όλες τις, τις προσπάθειες. Γιατί το θέμα αυτό ήταν περίπλοκο, αλλά και απ' την άλλη πάρα πολύ αναγκαίο. Και μιλώ για το τέταρτο πακέτο για τους ιδρώμου. Και μετά την πρώτη φάση μπόρεσαν να επεξεργαστούν όλα αυτά τα περίπλοκα νομοθετήματα. Να φιλουθεί η κατάσταση, για να υπάρχει μια συνέπεια και συνοχή. Σχεδόν 100% επιτυχία. Βέβαια, λείπουν κάποια στοιχεία, κάποια στοιχεία τα οποία φαίνονται δευτερεύοντα, αλλά τελικά η κατεξοδότηση πράξης είναι τεχνοκρατικό θέμα και πάντως από ό,τι μας λένε ε, από την άλλη μεριά για τους κοινωνικούς εταίρους αυτά τα θέματα είναι καυτά. Βέβαια, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτική επιτυχία. Εγώ είμαι παλιά εδώ στο Κοινοβούλιο, ξέρετε, και ως ε, βουλευτήνα αλλά και ως ε, σύμβουλος για πολιτικά ζητήματα. Στις μεταφορές επομένως η τεχνική πλευρά χωρίς την πολιτική δεν κάνει τίποτα. Γιατί ακόμα έχουμε εκκρεμούσει διάφορες διαδικασίες επί παραβιάση κατά διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για του Οπότε, εάν δεν προχωρήσουμε και προς το πολιτικό μέτωπο, τότε θα ε, απονευρώσουμε τα τεχνικά θέματα που τα έχουμε προχωρήσει γιατί μιλάμε τώρα για πέμπτο, έκτο κλπ. πακέτο. Άρα θα πρέπει η επόμενη Προεδρία, η Λουξεμβουργιανή, να φροντίσει ούτω ώστε κάτι να γίνει και όσον αφορά τον πολιτικό πυλώνα. Εσείς, ακόμα και μετά την Προεδρία σας, μπορείτε να βοηθήσετε γιατί ξέρετε το θέμα. Να σας ευχαριστήσω επίσης και για τα σχετικά όψαν και οι συνάδελφοι αφορούν τις στατικές επενδύσεις. Θέλουμε μεταξύ μεταφοράς, προϋπολογισμού, ε, καλύτερη συνεργασία. Αυτό αφορά και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η ευαισθησία που έχουμε για τέτοια θέματα θα πρέπει να μεταφερθεί σε έργα. Έχουμε αυτές τις περικοπές ενώντας εκατομμυρίων που υπέστησαν οι μεταφορές. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση των επιδοτήσεων. Είναι κάτι σημαντικό και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί για το Γεβραλτάρ Εμείς το βλέπουμε σαν θέμα διμερές. Δεν τα θυμάται καλά η κυρία Φώστερ που είπε ότι το ρύθμισε η κυρία Λογιόλα το Παλάθιο όχι, όχι. Γιατί ήταν πάντα θέμα αυτό με τις κυβερνήσεις της δεξιάς. Το εκμεταλλευόντουσαν ε, πολιτικά και ο κύριος Μωρατίνος ε, έκλεισε τη συμφωνία της Κόρδοβα. Στη συνέχεια είχαμε κάποιες παραβιάσεις όμως. Για την υφαλοκρηπίδα εκεί. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα και σε σχέση με τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Είναι διμέρες το θέμα, αλλά θα πρέπει να επιληθεί. Ρώσον αφορά τη διάσκεψη για τις μεταφορές, είναι πολύ ευχάριστο ότι εσείς ε, βοηθήσατε την Επιτροπή και την Επίτροπο Μπούλτς γιατί καθώς υπάρχει το κομμάτι το δημοσιονομικό το κομμάτι το κοινωνικό. Τι θα γίνει δηλαδή με τους εργαζόμενους στις μεταφορές στο άμεσο μέλλον, τότε που θα προκύψουν τα πραγματικά προβλήματα. Πώς θα τους ενσωματώσουμε στους διάφορους κλάδους και τομείς. Οπότε και εσείς θα πρέπει στο μέλλον να στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εμφαθύνουμε στο τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση, με τους εργαζόμενους, όσον αφορά την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Ο Πρόεδρος. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω την Λετωνική Προεδρία για τη δουλειά που έχει κάνει στο τέταρτο πακέτο. Είναι ένας φάκελος ο οποίος πραγματικά χρειάστηκε, μας αφαίρεσε ώρες ύπνου. Αλλά πραγματικά κάνατε πολλές προσπάθειες, πολύ σοβαρές και θα ήθελα να σας πω με ειλικρίνεια πως δεν αξίζατε να περάσετε αυτά που περνάτε τώρα με τις προθεσμίες και με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πραγματικά δεν το αξίζατε. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε μια συμφωνία και να μπορέσετε να κλείσετε εσείς την Προεδρία σας με τα θέματα αυτά τελειωμένα. Το λέω με ειλικρίνεια. Και ελπίζω πως το Συμβούλιο θα κινηθεί λίγο προς την πλευρά μας. Τώρα να σας πω πως σήμερα μου τηλεφώνησαν κάποιοι εκπρόσωποι του κλάδου που τόσες πολλές προσδοκίες έχουν από τη δική μας έκθεση, τουλάχιστον για το τεχνικό πυλώνα και μου είπαν πως ανησυχούν και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν είναι πως Θέλουν να εμφανιστεί επιτέλους αυτοί αυτός ο τεχνικός πυλώνας και δεν μπορούν άλλες καθυστερήσεις. Και δεν καταλαβαίνουν, βιάζεται ή όχι να το εγκρίνει το τεχνικό κομμάτι το Συμβούλιο, γιατί το άτομο που μου τηλεφώνησε, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό κλάδο για την Ευρώπη, δεν ήξερε αν το Συμβούλιο θα δώσει και μία προθεσμία πέντε ετών για την εφαρμογή. Αυτό δεν το γνώριζαν. Γιατί το να βιάζεται κάποιος και να ανησυχεί κάποιος πολύ για το να δώσει απόκριση στον κλάδο, τότε αυτός θα πρέπει να προσπαθήσει και με τις προθεσμίες. Έτσι ώστε η οδηγία αυτή, αν καταλήξει σε κάποιο αίσιο λιμάνι, να εφαρμοστεί και να μπει στη το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους είναι ένα πακέτο το οποίο αποτελείται από δύο πυλώνες, τεχνικό και πολιτικό. Και όπως είπαν και κάποιοι συναδελφοί, αν ακολουθήσουμε αυτό το επιχείρημα για το ότι πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να εφαρμοστεί το τεχνικό σκέλος, όταν εσείς αφήσετε την Προεδρία στο Λουξεμβούργο, βοηθήστε τους, βοηθήστε τους να πετύχουν ένα συμβιβασμό στο Λουξεμβούργο. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την κοινωνική διάσταση του θέματος. Γιατί αν μέσω του πακέτου αυτού και μέσω της συζήτηση αυτής δεν προχωρήσουμε στο θέμα της διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών μεταφορών, που αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τότε εδώ το πακέτο, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να δούμε και τα κοινωνικά θέματα, μια και είμαστε τη στιγμή που χρειάζεται η καινοτομία, που χρειάζεται να δημιουργήσουμε θέσεις ποιοτικέ απασχόλησης στον κλάδο αυτό, που είμαι σίγουρη πως θα δημιουργηθούν πιο εύκολα, εάν εμείς είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε με συνεπή τρόπο όλο το πακέτο σε όλη την Ευρώπη, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί. Και αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει μια έλλειψη σοβαρότητας, μια έλλειψη αυστηρότητας από όλα τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτό πια είναι ανεπίτρεπτο. Για τα δικαιώματα των επιβατών, να σας πω πως εγώ είμαι από τη χώρα των Βάσκων. Το Γεβραλτάλ, εμένα μου φαίνεται πως αποτελεί μια πρόφαση που χρησιμοποιείται για να μην προοδεύσουμε στο θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών. Και αν το ζητήσει το Συμβούλιο ως μήνυμα, καλό θα είναι να πούμε πως πρέπει να πιέσουμε τα δύο κράτη για να συμφωνήσουν στο θέμα και να χρησιμοποιήσουν αυτή την πίεση που υπάρχει μέσα σε τούτο το φάκελο για να ζητήσουμε από αυτά τα δύο κράτη να συμφωνήσουν γιατί σε άλλους φακέλους που ενδιαφέρεστε πιέζετε. Και γι' αυτό σας παρακαλώ και εδώ να απεμπλακεί το θέμα αυτό που είναι πολιτικό και ζητώ από την Προεδρία της Λατωνίας να κάνει μια τελευταία προσπάθεια ε, μέχρι το τέλος της Προεδρίας της. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να μιλήσω σε σχέση με το σχέδιο Juncker φαίνεται να είναι ένα σχέδιο προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, η ανάκα, να έρθει η ανάκαμψη στην Ευρώπη. Βλέπω όμως ότι το Συμβούλιο ε, παίρνει τα χρήματα και τελικά δεν τα αξιοποιεί όπως πρέπει. Αυτό είναι άδικο. Και το δεύτερο που είπε ο κύριος Σερτού, ο Horizon 2020 είχε 70 δις. Το Connecting Europe 26 δις. Όμως θα δώσουμε πιο πολλά λεφτά από όσα έχει το ορίζον 2020. Δεν έχει καμία λογική και δεν την αντιλαμβάνεται κανεί τη λογική μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Ιδιαίτερα καθώ έχουμε περάσει και δύο χρόνια να μελετάμε και να προωθούμε ευρωπαϊκά έργα και σχέδια, τα οποία θα εξυπηρετούσαν, τα οποία είναι έτοιμα και τα οποία τώρα εξετερώνονται και ακυρώνονται. Από αυτά τα σχέδια θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οδικές, οδικούς άξονες κάπου. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το τι θα γίνουν τώρα αυτά τα λεφτά και αυτά τα σχέδια. Ποιο, ποιο έργο θα προωθηθεί δηλαδή. Επίσης ξέρουμε ότι με, το, με τις συνθήκες Λισαβόνης ε, αυτά τα μεγάλα σχέδια έχουν πολύ μεγάλη σημασία και, και για την χειραφέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμω το Συμβούλιο και η Επιτροπή θέλουν να χειραγωγήσουν το Κοινοβουλίο και να παίρνουν τι αποφάσει. Εμεί, ω συγκητέ, καταφέραμε με τι κατεξουσιοδότησης πράξη να υπάρχει αυτή η ίδια συζήτηση, η παραλαμβανόμενη όπως και με το σιδηροδρομικό πακέτο. Αρχίσαμε να συζητούμε και να βρίσκουμε συμβαστικές λύσεις με τις νομικές υπηρεσίες. Τρία όμως προκύπτουν ως ιδιαίτερα προσκόμματα για τις κατεξιδότησης ε, πράξεις Υποτίθεται ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα τεχνολογικά, τεχνικά, νομοτεχνικά ζητήματα και εκεί μπορεί να τα αναλαμβάνει η Επιτροπή μόνο, αλλά σε ορισμένα ζητήματα πρέπει και εμεί να είμαστε θέση να τοποθετηθούμε. Και εδώ έρχεται το μήλον τη έρευνα. Είτε πρόκειται για σχέδιο Juncker, είτε για οτιδήποτε άλλο, οι κάτι εξουδότηση συμπράξει πρέπει να μην παραβιάζουν το πρωτογενές δίκαιο του Κοινοβουλίου ως νομοθέτη. Δεν μπορεί να το παραβιάζουν, όπως και με σιδηροδρόμους. Βλέπω όμως ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές προσπάθησαν, απέτυχαν και πολλές φορές έγιναν και προσφυγές στο δικαστήριο που καθυστέρησαν πολύ. Λοιπόν, το delegated acts είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Δεύτερον, προθεσμίες, χρονοδιάγραμμα. Πέντε χρόνια θέλει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή έλεγε ένα έτος, ε, δύο έτη, λέγαμε ένα. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη είτε μπορούν να πάνε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Γιατί όμως πρέπει να περιμένουν πέντε χρόνια μέχρι να υλοποιηθούν. Ας διαλέξουν μέσα δύο χρόνια. Ο κόσμος περιμένει, ο κλάδος περιμένει να υπάρξει επιτέλους μια κοινοτική, μια ευρωπαϊκή αξία κοινή με μια ευρωπαϊκή απόφαση. Και τρίτο σημείο, το σύστημα ασφάλειας στους Έχουμε πολύ δυσάρεστη και κακές εμπειρίες τελευταία 10 χρόνια με 10.000 ε, χιλιόμετρα που όμως δεν καλύπτουν, ε, δεν μπορούν να καλυφθούν από έναν σειρμό. 10.000 χιλιόμετρα έχουν αυτό το σύστημα ασφαλείας, αλλά δεν μπορεί να τα καλύψει ένας ενιαίος σειρμός. Τώρα βλέπουμε ότι πάει να πάρει και άλλη καθυστέρηση αυτή η υπόθεση. Δηλαδή και πιο πολύ χρόνο και πιο πολύ χρήμα θα κοστίσει όλη αυτή η υπόθεση λόγω της ε, παράτασης. Πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία. Με την ε, υπηρεσία των σιδηροδρόμων την ΕΡΑ πρέπει να βρούμε μία λύση. Έχουμε ένα συντονιστή, τον ΦΙΝΚ ο οποίο 10 χρόνια τώρα ασχολείται με την υπόθεση αυτή. Κάθε φορά που τον ρωτάμε μα λέει τα πράγματα είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι αυτά τα τρία πράγματα τα οποία θεωρούμε απαράδεκτα και σα παρακαλούμε. Και βεβαίω έχω κάθε έπαινο να εκφράσω για εσά, την Προεδρία σα και για του συνεργάτε σα που βρίσκονται στο πίσω, στα πίσω έδρανα. Πρέπει όμω να εξασφαλιστεί και μία λύση συνενετική για τους τρεις αυτούς τομείς έχει κάνει πολλές ε, παραχωρήσεις στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. Ε, τώρα έχει έρθει η ώρα να κινηθεί και το Συμβούλιο. Ο κύριος Φαντενκάμπ είπε ότι την περίφημη φράση από το τέλο μακάριζε» όπως λέμε εμείς ε, στα γερμανικά πριν κλείσει η μέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλή. Ε, λοιπόν, ελπίζω στις μέρες που σας έχουν μείνει ακόμα να τα καταφέρετε Μεγάλη πρόκληση, χρειάζεται συμβασμός πάντως. Και δεν νομίζω ότι μπορείτε να είσαστε απόλυτα ικανοποιημένος αν αυτά τα τρία ζητήματα δεν έχουν ρυθμιστεί. Πάντως η επικοινωνία και η, ε, το επίπεδο επικοινωνίας μας ήταν πολύ καλό και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ τώρα να λάβετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γράμμα, λέει ο Υπουργός αγαπητοι βουλευτέ, βουλευτές, πρώτα-πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ. Επικοδομητική ήταν η συνεργασία μαζί σα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όλα αυτά που είπατε για την Λεδονική Προεδρία. Οφείλω να πω ότι τον Ιανουάριο που συναντηθήκαμε, ανλάβαμε κάποιες δεσμεύσει. Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα τηρήσουμε όσο γινόταν πιο ολοκληρωμένα. Βέβαια. Για να σα πω τώρα πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τι εσωτερικέ πρωτέ οδού, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ζήτημα. Προσπαθήσαμε να θεσπίσουμε ενιαία κριτήρια. Την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο καταλήξαμε σε συμφωνία. Κατά 90% καλύφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η επομένη Προεδρία πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει την συμφωνία μαζί σας για αυτό τον τομέα που είναι τόσο σημαντικός. Τώρα, όσον αφορά τη δεσμή μέτρων για τους αεροδρόμους, υποσχεθήκαμε να προωθήσουμε και τον τεχνικό πυλώνα και τον πολιτικό. Εντάξει, για τον πρώτο πυλώνα προχωρήσαμε ταχύτερα. Αλλά όσον αφορά τώρα τον δεύτερο τον πολιτικό πυλώνα αφιερώσαμε πολλή ενέργεια προσπαθήσαμε πολύ νομίζω ότι λίγα θέματα εκκρεμούν ακόμη και η Λουξεμβουργιανή Προεδρία ανέλαβε να καταλήξει σε συμφωνία τον Οκτώβριο που θα υπάρξει η Υπουργική Σύνοδος νομίζω ότι το θέμα θα προωθηθεί αρκετά γρήγορα θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό για τις υποδομές, τη σχετική διαχείριση, για την διακυβέρνηση. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Και σε άλλα θέματα προχωρήσαμε, αλλά πάντως ειδικά για τον πολιτικό πυλώνα, σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να καταλήξουμε σε κάποιους συμβασμούς. προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ευέλικτοι. Οι φορμαστικές πράξεις για την εξοδότηση πράξης, εδώ ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά και εδώ θέλαμε να επιληθούν τα προβλήματα. όχι μόνο για να καυχηθούμε ότι και αυτό το καταφέραμε, αλλά γιατί η ευρωπαϊκή βιομηχανία περιμένει πώς και πώς να δοθεί κάποια λύση. Αλλά και οι Ευρωπαίοι πρόκειται να ωφεληθούν αν εκεί προχωρήσουν. Άρα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τις τελευταίες εβδομάδες προεδρίας μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και στην αεροπλοεία είχαμε σημαντικά προβλήματα. σημαντική υπόθεση και αυτή για όλη την Ευρώπη. Και ξέρουμε ότι και εδώ προχωρήσαμε αρκετά γρήγορα. Αλλά χάσαμε ακόμα τις αγοράς σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Άρα θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό και την σχετική Υπουργική Σύνοδο όσον αφορά την πολιτική αεροπορία. θέλαμε να δούμε πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και επίσης συζητήσαμε σε εκείνη την σύνοδο διάφορα νομοθετικά ζητήματα. Σχεδόν λύθηκαν όλα τα προβλήματα όσον τα δικαιώματα των επιβατών. Κρεμούν κάποια ζητήματα ακόμη Και όσον αφορά το ζήτημα του Γιβραλτάρ, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί δεν ήταν τόσο δύσκολο, θα είχε επιληθεί πολύ καιρό τώρα. Ελπίζουμε να κάτι να γίνει για να προχωρήσουμε. Τεχνικού χαρακτήρα συμβασμοί έχουν επιτευχθεί σε πολλά μέτωπα. Να, ας πούμε, ε, τα μη πατρωμένα ε, αεροσκάφη, Πρόκειται για ένα νέο τομέα. Θα πρέπει να είναι πρωτοπόρα η Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Έχουμε επίσης και την ε, δήλωση της Ρήκας. Είπαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πολλές κατευθύνσεις ε, ασφάλεια, τεχνικά ζητήματα, ε, κοινά πρότυπα, γιατί εάν δεν μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτά τα κοινά πρότυπα, τότε κάποιο άλλος θα το καταφέρει. Αλλού. Οπότε και τότε θα έχει χαθεί η μάχη. Γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε, γι' αυτό και βάλαμε αυτό το θέμα σαν προτεραιότητα. Τώρα, οδική ασφάλεια. Πρέπει να σας αναφέρω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Για την Ευρώπη, ε, στην Υπουργική Σύνοδο Ακούσαμε την εισήγηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το φθινόπωρο θα υπάρξει μια άλλη έκθεση πιο συγκεκριμένη. Πάντως πρέπει να σας πω ότι οι αμέσως επόμενες προεδρίες οι οδικές φορές της πόλης θα είναι θέμα μεγάλης ψηλής προτεραιότητας. Θα καθορίσουμε στόχους και θα βελτιωθεί επομένως η ειδική ασφάλεια. Τώρα, στρατηγικές επενδύσεις. Προσφέρονται ευκαιρίε για τις μεταφορές από το ΕΦΣΙ. Έτσι θα έχουμε χρηματοδότηση μεγάλων ε, έργων και σχεδίων που θα αφορούν τις μεταφορές και τις υποδομές. Θα γίνει μεταφορές πιο ανταγωνιστικές. Το αναφέρατε κι εσείς για τα προγράμματα τα οποία θα είναι το κλειδί για το μέλλον των μεταφορών. Είμαι πεπισμένος ότι όλα αυτά τα μέσα που διαθεσή μας θα τα προσαρμόσουμε ε, στις ε, ανάγκες του, του κλάδου των μεταφορών να αναπτυχθεί περισσότερο. Τώρα όσον αφορά το γενικό dumping για τις μεταφορές. Και αυτό το θέμα συζητήθηκε στο Συμβούλιο όταν συζητήσαμε για τις οδικές μεταφορές. Όταν συζητήσαμε το πώς θα ρυθμίσουμε τις οδικές μεταφορές με βαρέα οχήματα. Αλλά τα συζητήσαμε και για τις ε, αεροπορικές μεταφορές. Συζητήσαμε θέματα dumping. διευνήσαμε πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποιες κοινέ αρχές. Και για μισθούς και αμοιβέ εργασία. Νομίζω με αυτά τα ζητήματα θα ασχοληθούν και οι επόμενες πρόεδρες. Τώρα για τα διευρωπαϊκά δίκαια, δίκτυα μεταφορών, είναι και 30 Ιουνίου, θα έχουμε 1.200 πρόσωπα που θα έρθουν να συμμετάχουν στις σχετικές μέρες εορτασμού ε, αυτών των δικτύων. Θα εξετάσουμε επομένως ε, τι θα γίνει με τους σχετικούς διαδρόμους αυτών των διευρωπαϊκών δικτύων θεωρούμε ότι θα μάθουμε πληροφορίες θα έχουμε για αυτά τα δίκτυα τι θα γίνει με την Βαλτική με το διάδρομο στη Βαλτική εμείς αυτό θα το προωθήσουμε για την περιοχή εκείνη είναι πολύ σημαντικό το έργο θα πρέπει οι βαλτικές χώρες και αυτές να ενταχθούν σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο του σύμπαν. Πρόκειται για ρεκόρ επένδυση ε, κάποιου έργου στην περιοχή της Βαλτικής. Επίσης κάποιοι με ρωτήσατε τι, πώς συνεργαστήκαμε με τις παλαιότερες προεδρίες, πώς θα συνεργαστούμε με τις επόμενες. Εμείς είχαμε στάση ενεργητική, δυναμική, προς όλες τις κατευθύνσεις προσπαθήσαμε να συμβαστούμε όπου ήταν δυνατόν. Έχουμε στενή συνεργασία και θα έχουμε με την Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Το ίδιο ίσχυσε και με την ε, Ολλανδική Προεδρία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε αυτό το εξάμεινο. Είμαστε μικρή χώρα, αλλά αφιερώσαμε ό,τι πόρους μπορούσαμε για να προωθηθούν θέματα σημαντικά για την Ευρώπη. Πάντως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κράμερ, τους εισηγητές, τους και εισηγητές για τη βοήθειά τους. Ελπίζω να συνεχίσει η συνεργασία μας και ελπίζω τελικά θα συμβαστούμε όσον αφορά τα νομοθετήματα για τους υδροδρόμους. Ο πρόεδρος. Bei so viel Beifall Περιπτώσει χειροκροτήματα δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμω, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για τον απολογισμό αυτή τη πρώτη σα Προεδρία για τη Λετωνία. Ευχαριστούμε πολύ και για τη δουλειά σα και για τι απαντήσει που δώσατε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ. Καλή επάνωδο. Και φυσικά θα παραμείνουμε σε επαφή. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Νέες προκλήσεις για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη. Η Σαμπέλα Λεμόντε είναι η συγγετρία. Καθυστέρησε το αεροπλάνο της. Γνωστά φαινόμενα. Αλλά ήρθε το μεταξύ. Η Σαμπέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θεωρώ ότι όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και τα αεροδρόμια υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε ακόμη. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης που αναδεικνύουν το πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την οικονομία μας, για την Ευρώπη, πολύ σημαντικό. Αλλά είναι σημαντικό και για την ΜΜΕ, για την απασχόληση των νέων και των γυναικών. Και την επόμενη δεκαετία προβλέπεται αύξηση περίπου 140 εκατομμυρίων τουριστών που θα έχουν ως προορισμό την Ευρώπη. Αυτό θα είναι διεθνέ φαινόμενο από παντού δηλαδή, οπότε έχει σημασία και αυτή μας η πρόταση. Θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, θα πρέπει να γίνει περισσότερα για τον υπεύθυνο βιώσιμο τουρισμό. Θα πρέπει όμως να δούμε και τι γίνεται και για κάποια άλλα ζητήματα που είναι της καυτής χειρότητας. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι το πώς θα παραμείνουμε ο πρώτος παγκόσμιος προορισμός. Ε, βέβαια ε, αυτό δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν και άλλοι ε, προορισμοί που ανεβαίνουν. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα. Εξελίσσεται πολύ γρήγορα ο τουρισμός αλλά θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις οι οποίες είναι καταιγιστικές. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους στόχους που έχουν τεθεί, ε, και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι σχετικέ προκλήσει. θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πλευρά ε, οικονομική, τι γίνεται με του πόρου που έχουμε που είναι κυρίω διαρθρωτικοί, ε, να δούμε τι γίνεται και με τι μελέτε επιπτώσεων, να δούμε πώ θα είναι καλύτερη η λειτουργική στρατηγική μα σε σχέση με τόσα όσα θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι στρατηγικό ο τομέα αυτό. άρα θα πρέπει να έχουμε συνέπεια και συνέχεια. Δεύτερον, θέμα. Έχουμε διάφορους υποτομείς που υπάγονται στον τουρισμό, δηλαδή γιατί έχει εγκάρσιο χαρακτήρα, οριζόντιο χαρακτήρα, οπότε όλα αυτά τα θίγουμε στο κείμενό μας και γι' αυτό νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να εστιάσουμε προσοχή μας σε μερικά από αυτά τα ζητήματα, αυτά που τα θεωρούμε στρατηγική σημασία. Άρα, τι θα γίνει με με την Ευρώπη ως προορισμό και αυτό να λάβει το χαρακτήρα ενός εμπορικού σήματος. Αυτό πρέπει να το τα κρατημέλια, πρέπει να βοηθηθούν. Άρα να διευκολυνθεί η συνεργασία. Συνεργασία κράτους και ιδιωτικοτομία. Να δούμε τα νέα προϊόντα διεθνούς χαρακτήρα, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, μια στρατηγική μακροπεριφερειακή. Να δούμε πώς θα ξεφύγει από τον εποχιακό χαρακτήρα ο τουρισμός. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποια προϊόντα, τα οποία να στοχεύουν σε ηλικιακές ομάδες πληθυσμού. Ηλικιωμένους, νέους. Άρα να υπάρξει σχετική κατάρτιση, ενημέρωση των καταναλωτών, Επίσης, βιώσιμος τουρισμός και υπεύθυνο τουρισμός. Εδώ έχουμε τους προορισμούς αριστείας. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα ευφύα σύστημα. Θα πρέπει ο τουρισμός να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, στην βιοπικιλότητα, στις ορεινές περιοχές, αλλά και στις παρακτήσεις. και θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει επίσης και με τις ε, διαδρομές κατάλληλες για ποδήλατα. Άρα, κινούμαστε τώρα στο περιβάλλον της οικονομίας του διαμοιρασμού, share economy. Αυτό μας απασχόλησε και στην ακρόαση. Και επίσης είναι επίκαιρο με την ευκαιρία της έκθεσης Expo στην Ιταλία. Υπάρχει ζήτηση και θα πρέπει να καλυφθεί. να αξιοποιήσουμε τις ιδιομορφίες του κάθε τόπου, να προσαρμοστεί ο τουρισμός στις, ε, στα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, να δούμε τι θα γίνει με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά το πόσο δόκιμη είναι κάθε ενέργεια και να υπάρχει κάποια επαγγελματική αντιμετώπιση. Όταν κάποια δραστηριότητα έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, ε, τότε θα πρέπει να διέπεται από την νομοθεσία όπως γίνεται με όλους τους κλάδους. Αυτό έχει και τη φορολογική πτυχή, γιατί πρόκειται για κάποιο είδους ε, ε, δραστηριότητα που παράγει κέρδος και άρα υπόκειται σε φορολογία. Να αξιολογηθεί επομένως το θέμα της οικονομικής επίπτωσης. γιατί εδώ πέρα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το θέμα το, του, του κέρδους, των εσόδων από, την, από τον τουρισμό. Να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την πρόσβαση στα διάφορα δίκτυα. Εκεί που τουρίστας ε, στο ίντερνετ ψάχνει ε, που θα κάνει διακοπές, αλλά ε, υπάρχουν αδύνατα σημεία, δεν υπάρχει διαπροσβασιμότητα σε πολλά σημεία της αγοράς, αν θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των tour operators με τις επιχειρήσεις που κινούνται στο ίντερνετ και έτσι να είναι πιο αποδοτική αυτή η μέθοδος. Και αυτό να καλυφθεί και με προγράμματα ευρωπαϊκά χρηματοδότησης. Μιλούμε για ψηφιοποίηση όσον αφορά τα εισιτήρια, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ αναγκαίο να γίνει και αυτό έχει βέβαια να κάνει και με το κατά πόσον υπάρχει Wi-Fi ασύρματο Ιντερνετ ε, δωρεάν ή κατά πόσον υπάρχει ε, φτηνή περιαγωγή και φυσικά πρέπει να καλυφθούν και οι περιοχές της υπαίθρου πιο δυσπρόσθετε όπως τα βουνά οπότε να βελτιωθεί η επίδοση που έχουμε σήμερα όσον αφορά την προσβασιμότητα στα τρένα γιατί δεν είναι αρκετή το τρένο. Και δεν μιλώ μόνο για την προσβασιμότητα από τους αναπήρους, αλλά και για άλλε δυσκολίε που έχει κάποιο κόσμος. Μπορεί να είναι και εποχιακού ή προσωρινού χαρακτήρα. Άρα αυτό προσφέρει μία ευκαιρία. Και αυτή η ευκαιρία δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από την Αδράνη. Όταν τώρα κάποια τελεία για να μιλήσουμε και οι άλλοι συνάδελφοι και βεβαίως ε, είμαι πρόθυμη να καλύψω όλες τις ε, προτάσεις για το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και πιστεύω ότι μπορούμε να καλύψουμε τις απόψεις. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πριν προχωρήσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών του κυρίου Φλέκενστάιν, 18 μέλη της European Transport Workers Federation, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές. Καλώς ήρθατε. Έχουμε μια κάποια πίεση χρόνου εδώ μεταξύ και παρακαλώ οι σκιώδεις ηγητές να μην μιλήσουν τώρα από δύο λεπτά έκαστος. Κυρία Μοντερό Αγγία. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική προσπάθεια που έχει κάνει και για το γεγονός πως έχει εντάξει σημεία πολύ σημαντικά, διαφορετικά από ό,τι συζητάμε συνήθως. Ψηφιοποίηση, η συμμετοχική η οικονομία, η οικονομία του διαμοιρασμού κτλ. Σημεία τα οποία είναι πολύ σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση. Και τώρα, μιλάμε για τον τουρισμό, το θαλάσσιο και τον παράκτιο. Νομίζω ότι για τη γαλάζια οικονομία είναι από τα πιο ουσιαστικά, όπως είπε και η συγγήτρια. Και πρέπει να δούμε ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οι συγκεκριμένοι στόχοι για τον παράκτιο και το θαλάσσιο τουρισμό. Τρία εκατομμύρια Τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι αποσχολούνται στον κλάδο αυτό και άλλα πολλά εκατομμύρια εργαζόμενοι συνδέονται με, την, με τον παράκτη τουρισμό. Σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα και στα διάφορα τουριστικά πακέτα που είναι η υπηρεσίες αναψυχής στη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ, γαστρονομικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός κτλ. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, να φτάσει σε απόμακρα μέρη. Θα πρέπει να είναι πιο εύκολη, για παράδειγμα, η χορήγηση θεώρησης, να μην υπάρχουν εμπόδια ε, στην ε, επίσκεψη από ε, ξένους τουρίστες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρακολουθήσουν ε, τι γίνεται στις ε, περιοχές αυτές και να κάνουμε ένα πανευρωπαϊκό διάλογο για να μοιραστούμε ε, τα συμπερίσματά μας και να έχουμε κάποια μακροπρόθεσμη συνεργασία. Όταν μιλάμε για παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη και το τι γίνεται με τις νησιωτικές περιοχές και κυρίως τις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές που υπάρχει πρόβλημα συγκοινωνιών και συγκοινωνιακής σύνδεσης. Πώς να αναπτυχθείς τουριστικά αν δεν έχεις επαρκείς συνδέσεις. Δεν θα πρέπει ο προπολογισμό μας να έχει μια συγκεκριμένη γραμμή που θα ε, περιχαρακωθεί για τα θέματα τουρισμού μήπως το εμπορικό σήμα του τουρισμού της Ευρώπης θα πρέπει να οριθεί εμπορικό όπλο και να συνδυαστεί με συγκεκριμένες στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να αναπτυχθεί. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν με την ε, χρηματοδότηση των θεμάτων αυτών από κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, Οπότε ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση και να επιτύχουμε ε, μια λύση που θα επιτρέψει στους πάντες να ταξιδεύουν χωρίς το κόμματα. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Λοτόφσκι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την έκθεση. Ο τουρισμός είναι βεβαίως ε, ιδιαίτερα σημαντικός τομέας σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να βρούμε λοιπόν λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να συνεχίσει να είναι ο υπαριθμόν ένα προορισμός για τους ε, τουρίστες, για τους επισκέπτες. Ε, δεν πρέπει βεβαίως να παραγνωρίσουμε εδώ τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, η καινοτομία. Είμαι όμως ακόμη επιφυλακτικο προς το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να αναλάβει δράση γρήγορα και να αντιδράσει γρήγορα στις εξελίξεις. Η γραφειοκρατία που έχει καταστεί συνώνυμη με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να αναλάβει μόνο συντονιστικό ρόλο και όχι νομοθετικό στην υπόθεση αυτή. Βεβαίως, σημαντικό θέμα είναι η προστασία του καταναλωτή. Υπάρχουν νέα μέσα, νέοι τρόποι προσφοράς υπηρεσιών που όμως μπορεί να οδηγήσουν και σε καταχρήσεις των δυνατοτήτων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να προκύπτουν και κυρίως σε θέματα φορολογικού δικαίου ε, καταστρατηγήσεις των ε, διατάξεων, των εθνικών διατάξεων. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ίδιες τις περιοχές στις οποίες επισκέπτεται ο ε, η νέα τεχνολογία, το διαδίκτυο μας επιτρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε οπουδήποτε στην Ευρώπη μια ε, περιοχή, έναν προορισμό, ακόμα και αν δεν είναι ο πιο ε, προβεβλημένος. Υπάρχουν ε, περιοχές στην Ήπεθρο, υπάρχουν μικρές πανσιόν, υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές που διατηρούν τις παραδόσεις τους, που επιτρέπουν στον τουρίστα να δει της, ε, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και όμως δεν είναι οι πιο προβεβλημένες. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε στον ιδιοκτήτη κάτοχο εκμεταλλευόμενο αυτή την, ε, ε αυτόν τον προορισμό του τουριστικό, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προβληθεί καλύτερα και ιδιαίτερα θέλω να σημειώσω ότι ε, πρέπει να γίνει σωστά, πιο σωστά τουλάχιστον η διατύπωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών όρων ότι αυτοί δεν μπορεί ποτέ να αξιοποιηθούν ως ε, μέσα, ως επιχειρήματα, ώστε να φέρουν μεταξύ ε, διαφόρων ε, περιοχών μια σχέση ανταγωνιστική, μια σχέση πολεμική. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ξεπεράσατε το χρόνο σας, Γιώργο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώντας τους φιλελεύθερους, θα ήθελα να στηρίξω την έκθεση αυτή και να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε για το σημαντικότατο αυτό ψήφισμα. Ο τουρισμός είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας και μας επιτρέπει να μοιραστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες γιατί είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και θα ήθελα στο εισαγωγικό τμήμα αυτής της ε, έκθεσης να αναφερθεί το πόσο θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο τουρισμός στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών σε όλο τον κόσμο. Στηρίζω ιδιαίτερα δύο σημεία της έκθεσης αυτής που αντιμετωπίζουν το νέο φαινόμενο της σύγχρονης οικονομίας και κυρίως του σύγχρονου τουρισμού που είναι η οικονομία του διαμοιρασμού. Θα ήθελα στην έκθεση αυτή να φανούμε πιο ανοιχτοί για, δυναμο... δυνατότητες που προσφέρει αυτή η... οικονομία του διαμοιρασμού, για το τι προσφέρει στην κλασική οικονομία και να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο ισορροπημένοι στο πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε έτσι ώστε να λειτουργήσει και αυτό το είδος η οικονομία προσφέροντας τις τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει. Δεύτερον, στηρίζω ιδιαίτερα την ψηφιοποίηση και τη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων στο θέμα του τουρισμού, συγκεντρώνοντας τα σχόλιά μου στην ευρυζωνικότητα και στο γεγονός πως είναι απαραίτητη αυτή για να χρησιμοποιήσουμε όλα όσα προσφέρει ο τουρισμός και κυρίως το να κλείσουμε την βυσαλίδα όχι μόνο στην κάλυψη την ευρυζωνική αλλά και στην ανάπτυξη των απομακρυσμένων νησιωτικών ε, ορεινών ή μειονεκτούσων περιοχών της Ευρώπης. Η κυρία Κιλόνεν. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι συντονίστρια. Και να σας πω ποιες είναι οι παρατηρήσεις από τον συνάδελφο που είναι σχεδόν συγητής που θα έπρεπε να πάει σε μια άλλη ε, συνεδρία και δεν μπορούσε να παραστεί. Θα καταλήξουμε σε ε, κάποιο ε, τελικό κείμενο από το σχέδιο κειμένου της κυρίας Δελμόντε όσον αφορά τον βιώσιμο τουρισμό, όσον αφορά τις, τις, τις προκλήσει αυτέ γιατί ο τουρισμό είναι πηγή κέρδου, πηγή σημαντική για την οικονομία της οπότε θα πρέπει να έχουμε καλύτερα πρότυπα και θα πρέπει επίση να υπάρξει σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων και συνθήκε εργασία, παρά το ότι από τον τουρισμό παράγεται το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίο χαρακτηρίζεται από τι πολύ βάρδες θέσεις Το σχέδιο κειμένου σα, αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη η πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον και η πολιτική ομάδα μα αυτό θέλει να προαγάγει τέτοιου τουρισμό. Επίση θέλουμε να είναι πιο προσβάσιμε οι υποδομές, οπότε και γι' αυτό έχουμε κατεβάσει κάποιε τροπολογίε για να διευκολύνουμε τους ε, αναπήρους να έχουν πρόσβαση στις ελληνικές. Τώρα όσον αφορά τους πόρους που διατίθεται για τον τουρισμό θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ενημέρωση, πληροφόρηση, ε, να διευκολύνουμε όλους του εμπλεκομένους όπως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους. Τελευταίο αλλά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την κατανομή των πόρων ε, στις τοπικές αρχές. Πρόεδρος. Κιθ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για άλλη μια φορά. Μέρο της G 11 που είναι για τους πράσινους η σκιώδη συγγήτρια. Και μάλλον βρίσκεται με τη δική σας σκιώδη συγγήτρια, λέει στην κυρία Πτυγκούε, ο κύριος Κιθ. Ε, σας ε, ευχαριστούμε κυρία συγγήτρια. Έχουμε πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε. κυρίω εκεί που ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι γίνεται με τη συλλογή των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τι στατιστικές του τουρισμού. Επίσης, ε, όπως λέτε, για την φυσική κληρονομιά, το περιβάλλον, ε, όλα αυτά είναι θησαυρός για δηλαδή το θησαυρό, όπω είπε η θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τι περιφερειακέ αρχέ και τα κράτη-μέλη να προαγάγουν τον οικολογικό τουρισμό. Και αυτό είναι υπόψη ε, από το κοινωτικό δίκαιο όσον αφορά τα διάφορα προϊόντα του τουρισμού. Έχουμε τις ακτές, έχουμε τα νησιά, έχουμε τα βουνά και όπως είπατε ε, πολλές περιοχές εκεί εξαρτώνται για τον τουρισμό, πρόσφατα κυρίως τον τουρισμό και έχουν πληγεί από την αλλαγή του κλίματος και γι' αυτό θεωρούμε πως η προστασία του κλίματος και η σχετική πολιτική θα πρέπει να διαπνέει κάποια ρύθμιση για μεταφορές, για ε, περιφερειακή πολιτική, για τουρισμό. Είναι τώρα για το θέμα του τουρισμού στις πόλεις. Θα πρέπει να δούμε το θέμα των μεταφορών προς και από το κέντρο. Θα πρέπει ε, αυτό να γίνει με τρόπο βιώσιμο και θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση που να ωφελεί και τους ε, κατοίκους και τους τουρίστες. Να υπάρξουν ε, για τον ήπιο τουρισμό κάποιο είδους πιστοποιητικά. Να γίνει κάποια ανάλυση κάποιων εκουσίων μέσων και έτσι να μπορέσουμε αυτές τις υπηρεσίες του ήπιου τουρισμού να τις αναδείξουμε. Να δούμε τι θα γίνει επίση και με το άλλο μας που έχουμε για τους προορισμούς αριστείας. Και ο κοινικός τουρισμός και ο ήπιος τουρισμός να βοηθηθεί από μέσα από τα δίκτυα που θέλουμε να οργανωθούν περισσότερο. Τέλος, θα πρέπει οι tour operators να προαγάγουν τα δίκτυα που χρησιμοποιούν τα, τα, τα ποδήλατα και οι ποδηλάτες, όπως ας πούμε το, τη διαδρομή εκείνη ε, του, του σιδηρού παραπετάσματος. Και επίσης θα δούμε τι θα γίνει με τα τρένα φλισταγήτως και με τα νυχτερινά τρένα, πρόεδρος. Κύριος ähm, zunächst einmal von meiner Seite an die Berichterstatterin. Ευχαριστούμε. Και εγώ λέω και Σαντού να ε, ευχαριστήσω τους συζητητέ και τους κοιόδες συγκεκριτές. Νομίζω ότι πολλά από τα σημαντικά ζητήματα και τα καθοριστική σημασία ζητήματα στον τουρισμό έχουν καλυφθεί. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερα διαφορετικά πράγματα να τονίσω. Απλώς θέλω να αφαιρθώ στο Branding Europe, να προβάλλουμε δηλαδή το σήμα Ευρώπη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στο τομέα ε, του τουρισμού ιδιαίτερως έχουμε να κάνουμε τεράστιο δυναμικό και νομίζω όλοι θέλουμε και μπορούμε να προβάλλουμε τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπον ενωμένο. Είμαστε μια περιφέρεια. Όταν έρχεται κάποιο από την Κίνα, από την από προ προς την Ευρώπη, δεν θέλει να δει μόνο ένα τόπο, θέλει να δει πολλέ περιοχέ. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το Branding Europe, να προβάλλουμε το σήμα τη Ευρώπη, δηλαδή. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ε, το θέμα της ψηφιοποίησης και της πρόσβασης σε διάφορα δίκτυα τηλεπικοινωνιών είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη. Ένα παράδειγμα, στη Βαλτική είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ εύκολο, πολύ συνηθισμένο να έχει κανείς σε δημόσια κτίρια, σε κτίρια δημόσιας πρόσβασης, ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε και αλλού. Και κάτι άλλο από την έκθεση Ουελή, Ένα ζήτημα σχετικό με την θεώρηση των διαβατηρίων. Εάν λάβουμε υπόψη ότι 1% των Κινέζων βγαίνει εκτός Κίνας για τις διακοπές του, αντιλαμβανόμαστε τι τεράστιο δυναμικό υπάρχει από τον τουρισμό και ίσως θα ήταν για λόγους τουρισμού να διευκολύνουμε τις διαδικασίες για θεώρηση βατήριων. Ευχαριστώ βέβαια και ιδιαίτερα την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ και να συγχαρώ και τη συνάδελφο κυρία Μόντε για μια εξαιρετική έκθεση για ένα κλάδο τόσο σημαντικό για την Ευρώπη που πολύ συχνά δεν την χάνει της απαραίτητης προσοχής ούτε σε επίπεδο προπολογισμού, ούτε σε επίπεδο επιμόρφωση και κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου, ούτε σε επίπεδο προώθησης και μάρκετινγκ στον υπόλοιπο κόσμο. Αν με επιτρέψετε, θα ήθελα να προσθέσω στα όσα υπόθηκαν. Έχουμε λοιπόν τα σημεία αριστείας στην Ευρώπη, αυτούς τους άριστους ε, τόπους. Είχαμε και ένα, πειρατικό, ένα πειραματικό πρόγραμμα που ήταν η πρωτοβουλία «Καλυψώ για τον κοινωνικό τουρισμό» με στόχο την προώθηση του τουρισμού ε, εκτός εποχής για άτομα τα οποία είτε γιατί οι χώρες τους δεν είχαν πρόσβαση σε κοινωνικό τουρισμό είτε γιατί ήταν τρίτη ηλικία είτε για κάποιους συγγενικούς δεσμούς αλλά εν πάση περιπτώσει ε, για κάποιους λόγους είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Βέβαια αυτό το πρόγραμμα δεν μακροημέρευσε και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει τι συνέβη με το θέμα αυτό. Είχε πολλές δυνατότητες. Έχει συμπεριληφθεί στην τρέχουσα στρατηγική για τον τουρισμό. Και τέλος να σας πω πως θα πρέπει να εντοπίσουμε και κάποιους τρόπους να γίνεται πιο ενδιαφέρον ο τουρισμός, ο περιπατητικός για παράδειγμα είμαι ο ποδηλατικός. Εμείς έχουμε ε, τη διαδρομή του Σαντιάγο Δε Κομποστέλα και αυτά να ε, συνδυάζονται με κάποιο είδους ε, πλαίσιο που θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έχουμε συνήθως αυτά τα είδη τουρισμού. Έχουμε και στο πακέτο για τις τουριστικές υπηρεσίες την ανάγκη να προσαρμόσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στις νέες συνθήκες. Και έχουμε και το τουρισμό και τις τρίτες χώρες εμείς ευνοούμαστε από το γεγονός πως άσχημο τουρισμό στην Τινησία, στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, όμως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιο είδους ανταλλαγές έτσι ώστε και εκεί ε, να ε, βελτιωθούν οι συνθήκες οι καθημερινές. Κύρκος. Ο κύριος Κύρκος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Ντεμόντε για την πολυσχεδή και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε αυτή την έκθεση και πολύ βιαστικά να τονίσω τρία σημεία το οποίο έχω βρει ιδιαίτερο ενδιαφέροντο. Το πρώτο είναι αυτό που καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση με κριτική εκτίμηση απόδοση των δράσεων του 2010. Αυτό είναι πολύ καλό να σχεδιάζουμε, αλλά πρέπει να επανερχόμαστε και να βλέπουμε και πώ αυτέ οι δράσει υλοποιήθηκαν ή όχι και τι μάθαμε από αυτέ. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό σήμα προορισμό Ευρώπη, ε, η συνεργασία του κράτους, ιδιωτικού τομέα, αλλά και η συνεργασία των κρατών για να καθορίσουμε τους όρους και επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το σήμα να μην ευτελιστεί, να είναι κάτι δηλαδή πάρα πολύ συγκεκριμένο και με μεγάλη αξία. Και το τρίτο είναι οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας που αναφέρονται, γιατί όντως μιλώντας για ένα ποιοτικό τουρισμό και αν θέλουμε να μεταβούμε σε ένα τέτοιο είδος τουρισμού, αυτό που θα το προσφέρει σίγουρα είναι η υψηλή ειδίκευση των εργαζομένων. Τώρα δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα, θα έβρισκα ίσω να υπάρχει μια αναφορά, όπως αναφερόμαστε στην πολιτιστική κληρονομιά και την βιοπικιλία, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στην πολιτισμική κληρονομιά, είναι το 40% του τουριστικού μας κίνητρου, η πολιτισμική κληρονομιά και ειδικά ε, όταν προσφέρεται υπεργαζόμενος υψηλής δεξιότητας αποκτά τεράστια σημασία στον τουρισμό μας και το δεύτερο είναι ο αγροτουρισμός, όχι μόνο ένα εκρηκτικά αναπτυσσόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά και ένας τρόπος που του ενισχύεται το πολλές φορές απελπιστικά χαμηλό εισόδημα των πραγματικών αγροτών. Με αυτό θα ήθελα να κλείσω και ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι την κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ, Τελίτσκα. Uh, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα συμφωνήσω με όσα υπόθηκαν από την ε, ομάδα μου. Θα ήθελα τώρα όμως να υπογραμμίσω κάτι που είπε η συγγήτρια. Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση της για την ε, ανάπτυξη του τουρισμού. Και εδώ επίσης θα με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονό ότι ε, μένεται ένας αγώνας για να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής για όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει να προχωρήσουμε. Και σε αυτό το βήμα δεν μπορούμε να μιλούμε για ψηφιοποίηση εάν δεν υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Θα πω και εγώ δύο λόγια, λέει ο Πρόεδρος κοινοτική διάσταση είναι βεβαίω την έχουμε. Έχουμε μια στρατηγική για τη Βαλτική, επί παραδείγματι. Τα κράτη που βρέχονται από τη Βαλτική θάλασσα έχουν κοινά σχέδια, τα προάγουν μαζί ε, και τα προβάλλουν από κοινού. Το ίδιο η στρατηγική για το Δούναβι. Με αυτό το πνεύμα νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και να ξεπερνάμε τα εθνικά σύνορα. Και αναφέρθηκε βέβαια ο τουρισμός ε, ο ποδηλατικός. Έχω κάνει την έρευνά μου. Είναι 44 δισεκατομμύρια ο κύκλος εργασιών του κύκλου εργασιών του ποδηλατικού ε, τουρισμού. Ε, ο ίδιος δηλαδή κύκλος εργασιών με αυτόν του τουρισμού της κρουαζιέρας. Εάν πάνε 44 δισεκατομμύρια στα λιμάνια δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά εάν μιλήσουμε για υποδομές ποδηλατοδρόμων, για τον ίσου δυναμικού ποδηλατικό τουρισμό, τότε κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά. Λοιπόν, πρέπει να τον προβάλλουμε. Είναι οικολογικά συμφέρον. Βεβαίω και την υγεία, κυρία Μάθημα. Μα βεβαίω και την υγεία μα. Πέντε χρόνια περισσότερο ζει ο ποδηλάτη από τον μη ποδηλάτη. Σα ευχαριστώ που με το θυμήσετε. Λοιπόν, έχει και οικολογικό αλλά και οικονομικό όφελο να προσφέρει πέραν τη υγεία. Και Κάτι άλλο. Επειδή πρέπει κάποιες περιοχές να διευρυθούν. Βαλτική θάλασσα που αναφέρθηκε παραδείγματι, η σεζόν, η τουριστική, μπορεί να είναι τρεις μήνες μόνο να αναφερθούμε στις διακοπές στη θάλασσα, αλλά αν Αν μεταστρέψουμε την τάση για τον ποδηλωτικό τουρισμό, τότε μπορεί να κρατήσει και δέκα μήνε τουριστική περίοδο στην Βαλτική. Κάτι άλλο όμω που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως ε, για το κατά πόσον θα διατεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για του ποδηλατοδρόμου. Εάν πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ποδηλατόδρομο σε μια πόλη κοντά κτλ., μπορεί να διατεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Άμα πω όμω ότι θέλω να κάνω τον ποδηλατόδρομο παράλληλα με την ακτογραμμή επί παραδείγματι, για να είναι καλό και για τον ε, τουρίστα ποδηλάτη, τότε θα πρέπει ίσω να εμπλακεί και η τοπική αρχή, η πόλη, γιατί βεβαίω κανένα ποδηλάτη δεν θέλει να ε, ποδηλατεί παράλληλα με έναν αυτοκινητόδρομο, Φερρυπίν θα είναι πολύ καλό να έχουμε γραμμέ παράλληλε, ο ποδηλατοδρόμο καλύτερα παράλληλους με τι ακτογραμμέ και τα ωραία, τα ωραία τοπία. Ευχαριστώ πολύ. Από την Επιτροπή θέλει κανεί το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' να ευχαριστήσουμε την κυρία Ντελμόντε. σε πολλά σημεία συμφωνούμε, όπως ε, το ότι θα πρέπει να προσέξουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των κοινωτικών πόρων το, όπως, ε, τους πόρους από το κόσμο, να γίνει κατάρτιση και εκπαίδευση, να δούμε τι γίνεται με την ψηφιοποίηση και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει πίσω σε σχέση με όσα έχει δεσμευτεί τον τουρισμό. Το αντίθετο. Θέλουμε να αξιοποιηθεί ο τουρισμό. Ο κλάδο είναι πολύ σημαντικό. Μόδα, ε, ε αγροτοδιατροφικά, ε, κατασκευές, ε, μεταφορές. Οπότε τώρα θέλουμε να προσέξουμε και την κοινοτομία και τα ψηφιακά και την κατάρτιση. Έχουμε επίσης τις ε, δημιουργικές προσπάθειες, τις πολιτικές προσπάθειες ούτως ώστε να συνδέσουμε αυτούς τους τομείς και με τον τουρισμό. Οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την προσέγγιση ότι πρόκειται για έναν τομέα που μέσα στους επόμενους μήνες ή χρόνια θα δημιουργήσει απασχόληση όχι μόνο στον Νότο, σε όλη την Ευρώπη και κυρίως για τους νέους. Αυτό είναι ο τουρισμός. Οπότε και σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να ε, βοηθήσουμε τον τουρισμό. Και θέλουμε να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο. Τώρα κάποια σημεία τα οποία ε, εθίγησαν και αναφέρθηκε και το όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί συμφωνούμε πρώτα πρώτα με το ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα τέτοιο σήμα που να αφορά την πρόθεση της Ευρώπης σαν τουριστικό προορισμό και όλες τι άλλες δράσεις που γίνονται από κράτη και από περιφέρειες να προωθήσουμε την Ευρώπη ας πούμε προ τους Κινέζους που ξέρουν ελάχιστα πράγματα για την Ευρώπη για το Παρίσι βλέπουν την Ευρώπη το ίδιο σαν ένα σύνολο πρέπει να του πούμε Όπω κάνουν οι Αμερικανοί πόσα επενδύουν στη, για την Αμερική ως προορισμό Μα το, και οι Ινδοί το ίδιο κάνουν ε, αφήνουν ένα σωρό λεφτά σε καμπάνιες τώρα ε, αυτό που είπαμε να αποσυνδεθεί ο τουρισμός από τον εποχιακό χαρακτήρα ε, και αυτό να καλύψει τους νέους και τους πιο ηλικιωμένους ε, αυτό θα είναι σημαντική απάντηση δεν πάνε μόνο οι, οι Κινέζοι και οι Βραζιλιάνοι οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον τουρισμό τον ποδηλατικό τουρισμό δώσαμε και εκεί προτεραιότητα επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό και οι διεθνωτικοί πόροι σε σχέση με τον τουρισμό λαμβάνουν υπόψη ε, το, θέμα το ενεργειακό. Άρα λιτώνουμε από εκπομπές και εξοικονομούμε ενέργεια με τέτοιου είδους τουρισμό όπως ο ποδηλατικός. Και βοηθούμε και στο στόχο Κατά καταπονήμηση αλλαγής του κλίματος. Τώρα, άλλη παρατήρηση. Θαλάσσιος τουρισμός. Όντως είναι σημαντικός τομέας. Έχουμε και μια ανακοίνωσή μας του 2014 και κάποιες δράσεις προτείνουμε πάνω σε αυτό. Η κυρία Αγιλάρ έκανε μια σωστή πρόταση για σεμινάριο, για συνάντηση με τους εμπλεκόμενους σε αυτόν τον τομέα. Σημαντικό. Άλλο. Διαφάνεια στην δαπάνηση των περιφερειακών πόρων για τον τουρισμό. Εμείς πρόκειται να συνέξουμε κάποια έκθεση όσον αφορά τους πόρους από το κόσμο και από τα περιφερειακά ταμεία όπως ξέρετε αυτά δεν διατίθενται με δική μας απόφαση αλλά αποφάσισε σε περιφερειακό επίπεδο πάντως οι αποφάσεις για τον τουρισμό βεβαίως και επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και κυρίως την απασχόληση για τις θεωρήσεις διαβατηρίων Συμφωνούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όπως γνωρίζετε, εμείς θέλουμε να υπάρξει απλούστευση του καθεστώτος και διευκολύνσεις. Και έχουμε εντυπωσιακέ μελέτες για το τι θα πει, τι επιπτώσεις έχει η απλούστευση του χαρακτήρα των ε, θεωρήσεων διαβατηρίων, ας πούμε για την Κίνα. Γι' αυτό που είπε η κυρία Πιλμπό όσον αφορά το καλύψω. Τονίζουμε ότι συνεχίζεται το κάλυψο, συνεχίζει να χρηματοδοτείται στα πλαίσια του κόσμου. Είναι προτεραιότητα για τον Επιτροπό μας. Μη σας τρώω άλλο χρόνο και καταχρούμε της υπομονή σας. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, εσύ παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρο Ευχαριστώ πραγματικά όλους τους και ηγητέ, τους συνάδελφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα ανέφεραν. Και μου φαίνεται πάρα πολύ ευχαριστώ ότι συμφωνούμε σε τόσα πολλά σημεία. Αλλά την άλλη μεριά ευχαρίστως να προσπαθήσω να τους καλύψω και να ανέβρω λύσεις για όλα όσα προτείναν θα πρέπει να εντάξουμε στο κείμενο ιδίως σας είπαμε στην αρχή όσον αφορά τον ε, παράκτιο τουρισμό, τον θαλάσσιο τουρισμό που είναι σημαντικός πολύ για την οικονομία που αφορά τον τουρισμό αλλά και κάτι θα πρέπει να γράψουμε και για τον πολιτιστικό τουρισμό. Άρα θα πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω που να είναι σαν χαρακτηριστικό της Ευρώπης ως προορισμού και να κάνει την διαφορά σε επίπεδο πολιτιστικό. Ακριβώς γι' αυτό μίλησα πριν για τον ε, τουρισμό πέρα από τα σύνορα, πώς θα υπάρχει κάποιο είδους ε, έλξη σε αυτό το επίπεδο, γι' αυτό είπα και για το εμπορικό σήμα ε, του προορισμού Ευρώπη και να λάβουμε υπόψη τις ιδιοτυπίες ε, του κάθε τόπου. Άρα θα πρέπει να μειώσουμε το, το, ευάλωτο των θέσεων εργασίας στον τουρισμό να υπάρχει μια συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση, να σταματήσει ο εποχιακός χαρακτήρας και η δουλειά στον τουρισμό να κρατάει όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στην χρονιά. Πολλοί είπαν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με την ψηφιοποίηση, να καταργηθούν τα έξοδα για την περιαγωγή. Αυτά να είναι προσφορές αυτονόητες για τον τουρίστα και Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα η καλομεταχείριση των ζώων. Να το λάβουμε υπόψη. Και για τον τουρισμό. Τέλος. Αρχή αρχή σας μίλησετε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την οικονομία. Βέβαια, διγλύτως κάποιος ο τομέας ε, από την κρίση σε σχέση με άλλους τομείς. Το εξαρτάται βέβαια από το μέρο, από το κράτο μέλος, αλλά ένα λόγο παραπάνω να μπορέσουμε να επενδύσουμε μακρόπνο. Και έτσι θα λειτουργήσει η οικονομία. Σα ευχαριστούμε και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τι τροπολογίε. Ευχαριστώ προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 24 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι. Μην το λησμονήσετε. Περνάω τώρα στο επόμενο θέμα τη ημέρα τη διάταξη, ευχαριστώντα φυσικά για μια φορά την εισηγήτρια και του κοιόδη εισηγητέ για τη συζήτηση. Επόμενο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Ε, λιμένες υπηρεσιών. Και μια και έχουμε εδώ κάποιους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα ακουστικά γιατί είναι όρθιοι. Θα τους καλέσω κατ' εξαίρεση σήμερα να καθίσουν και στα μπροστινά έδρανα για να μπορούν να παρακολουθούν την συζήτηση. Όλοι οι ακροατές μπορούν να πάρουν θέση όπου έχει ελεύθερες θέσεις. Ναι, φυσικά δεν με καταλάβατε στα γερμανικά, τα λέω και στα αγγλικά πάλι. Μπορείτε να καθίσετε στις ελεύθερε εδώ θέσεις για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις συνομιλίες στη γλώσσα σας ο καθένας. So, und wir Με μεγάλη αδημονία περιμένουμε την παρουσίαση στις προσωρινής εκθέσεως του Κνούτ Φλέκενστάιν. Όποιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω δύο λόγια για τη μεθοδολογία καταρχάς. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια έκθεση στην προηγούμενη θητεία με 500 42 τροπολογίες, 25 συμβαστικές προέκυψαν από αυτές και δεν μπορέσαμε καν να κλείσουμε το θέμα. Τις συμβαστικές στην έκθεσή μου τις λαμβάνω υπόψη μόνο εν μέρη. Εκεί όπου χρειάζεται θα τις ξανασυστήσουμε στις πραγματεύσεις. Δεν ήθελα όμως να γράψω συμβαστικές τροπολογίες εκ προημίου μέσα στο κείμενο για να μην χρειάζεται να κάνουμε συμβαστική πάνω στις συμβαστικές. Έχω λάβει γνώση της, ε, των θέσεων του Συμβουλίου σε ένα βαθμό της καταγράφω και αυτά στο κείμενο, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να καταγράψω αυτό που εμείς σκεφτόμαστε και να εξασφαλίσω έτσι ότι διαμορφώνουμε εμείς μια κοινή γραμμή για να προχωρήσουμε μετά σε μια κοινή γραμμή με το Συμβούλιο. Αυτό είναι η προσπάθειά μου είχα κάποιες επαφές και με τους εκπροσώπους των κατοχωρών στο θέμα αυτό. Κεφάλαιο 3 χρηματοοικονομική διαφάνεια και στο 4 διαβουλεύσεις ε, είναι τα κεφάλαια τα οποία λίγο πολύ έχω αντιγράψει την προηγούμενη έκθεση. Στο 2 έχουμε σημαντικές αλλαγές τις οποίες θέλω να σας αναφέρω, πρόσβαση στις αγορές ή μη πρόσβαση αγορά και ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και τις ε, χρηστές συνθήκες εργασίας, καλές συνθήκες εργασία. το τα πακέτα για τους λιμένες 1 και 2 προσπαθώ να, τους συμπερι, να τα συμπεριλάβω χωρίς όμως να ε, επιβαρύνω ή να προδικάζω την εξέλιξη το τρίτο πακέτο για τους λιμένες. Και τώρα πολύ στιγμό θα ήθελα να πω δύο λόγια στα επιμέρους σημεία. Πρόσβαση αγορές δεν είναι κομμάτι του κανονισμού πλέον, γι' αυτό αλλάζει τίτλο το κεφάλαιο και ονομάζεται πλέον οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών, διάφοροι τύποι οργάνωσης. Δεν θέλουμε να, υπο... Ε, να υπαγορεύσουμε κανένα ιδιαίτερο τύπο. Αφήνουμε στα κράτη-μέλη την ελευθερία να ορίσουν τον τύπο οργανωση των λιμένων του, τι είδου υπηρεσίε, πόσες υπηρεσίε κτλ. Αλλά μέχρι τώρα στο κεφάλαιο 2 δεν είχε εκφράσει κανείς την ικανοποίηση ότι, τα, ότι είναι επαρκές ε, και πλήρες ε, άλλοι λέγανε ότι περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, υπερβολικά πολλά στοιχεία, άλλοι λέγανε ότι δεν έχει αρκετά. Εξού και προχωρήσαμε σε αυτό το τρίτο πακέτο. Και χαίρομαι που μπορέσαμε με την Επίτροπο Μπύρους σε μια συνάντηση να συμφωνήσουμε ότι στο κεφάλαιο 3, χρηματοοικονομική διαφάνεια, ε, πρέπει να δοθεί και η έμφαση. Ε, επίσης, όλος ο κανονισμός έχει σαν στόχο τη βελτίωση της αγωνιστικότητας των κλειμένων. Για να βελτιωθεί όμως αυτή η ανταγωνιστικότητα πρέπει να μιλήσουμε και για ανταγωνιστικότητα, μάλλον για βελτίωση των εργασιακών συνθήκων και για κοινωνικό διάλογο. Θα φροντίσω ώστε να ανατραπεί η επιδείνωση των συνθήκων εργασίας και των θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους σε πολλούς λιμένες Ευρώπης. Έχουμε να κάνουμε πολύ συχνά με αποσπασμένη εργασία, με πολύ κακή κατάρτιση. Δεν μπορούμε στο 21ο αιώνα όμως να δεχόμαστε να έχουμε εργάτε του που πάνε στου τερματικού σταθμού και στέκονται στην ουρά περιμένοντα να βρουν δουλειά μόνο για τον επόμενο μήνα, Φερρυπίν. Στο κεφάλαιο 10 που γίνεται λόγο ε, για την λήψη υπόψη αυτών των συνθήκων από όλου του εμπλεκομένου. Ε, γίνεται λόγος επίση για την απαραίτητη κατάρτιση, κράτη-μέλη και εργαδοδότης, κοινωνικός διάλογος, ε, κατάρτιση προδιαγραφών ή επιπέδου συγκεκριμένων προδιαγραφών των ε, καταρτήσεων, ε, καλύτερες και ασφαλέστερες θέσεις εργασίας. Αυτά ζητούμε. Σαφές για μένα είναι ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα στον κανονισμό αυτόν. Αλλά ή μη τι άλλο μπορούμε να επισημάνουμε τα προβλήματα. Μπορούμε να πούμε ότι τα έχουμε βάλει στο στόχαστρο. Μπορούμε να πούμε ότι ε, μα ενδιαφέρει να συμβάλλουμε στην εξέβριση λύσεων. Τελευταίο σημείο, χρηματοοικονομική διαφάνεια, πυρήνα του κανονισμού και ιδιαίτερα σχέση με την συζήτηση σχετική με τις κρατικές επιχορηγήσεις. Η διαφάνεια λοιπόν ε, σε σχέση με τα κρατικά κονδύλια είναι ένα διαφιλονικούμενο ζήτημα. Όποτε γίνεται λόγος σε κρατικά κονδύλια ε, πάντα χρειάζεται να υπάρχει μια κάποια διαφάνεια σε επαρκή βαθμό. Ε, και εδώ έχουμε και τη σχετική τα σχετικά όρια για την αποζημίωση της επιστροφής των κονδυλίων. Πρέπει τα κριτήρια λοιπόν τα σχετικά για τις αποζημιώσεις να είναι διαφανή. Και λέω κριτήρια γιατί πρέπει τις διαπραγματεύσεις ανεξαρτήτως και αυτονόμως να τις διεξάγουν οι ίδιοι οι λιμένες. Η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό έχει πει στις προβλέψεις ότι μέχρι τα τέλη του 2015 μπορεί να έχει έτοιμη μια πρώτη, ένα πρώτο σκαρίφημα της αναθεώρησης του κανονισμού για τα block exceptions, για τις μαζικές δηλαδή Ε, μακάρι να τα καταφέρει. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να εκφράσει αυτές τις εξαιρέσεις. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με ένα κάποιο επίπεδο επενδύσεων ή μέχρι ενός επίπεδου επενδύσεις, αλλά και με, με επιχορηγήσεις που έχουν να κάνουν με ε, υποδομές και στις οποίες πρέπει να αναγνωριστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας. Ε, η αυτονομία επίσης των λιμένων. Υπάρχουν ε, κάποιοι λιμένες που μπορούν να προσφέρουν θέμενη αξία. Δεν είναι δηλαδή για μένα νοητό χρήματα τα οποία αφορούν τη Μαδρίτη να πηγαίνουν στην Βαρκελόνη τελικά αλλά να αξιοποιούνται τελευταία στιγμή για κάποια επαιτειακή εκδήλωση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των επιχορηγήσεων διαφάνεια όπως είπα, τίποτε το καινούριο ουσιαστικά αλλά ήθελα να πει οπωσδήποτε μέσα στο κείμενο. Και τελευταία παρατήρηση για την διαβούλευση με τους χρήστες και για την εποπτεία. Δεν υπάρχει λύση one size fits all που να καλύπτει δηλαδή όλες τις ανάγκες. Χρειάζεται μια ε, μετρημένη ε, διάταξη ή διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται διαβουλεύσεις με τους τελικούς χρήστες. Η μορφή όμως αυτών των διαβουλεύσεων θα πρέπει να ορίζεται από τους ίδιους τους λιμένες. Η δε εποπτεία σημαίνει μια ανεξάρτητη αρχή που θα πρέπει να ακολουθήσει έναν τύπο και αυτό θα το ορίσουν πάλι όχι εμείς αλλά τα κράτη-μέλη ε, θα ακολουθήσει τον τύπο ενδεχομένω του δικαστηρίου, του διευθυντικού δικαστηρίου, της αρχής διευθέτησης, της αρχής εποπτείας. Πάντως είναι μια λύση που μπορεί να είναι διαφορετική σε κάθε κράτος. Αυτά λοιπόν Ευχαριστώ πολύ τους αδέλφους που με βοήθησαν με τις αρχικές τους και προκατακτικές τους παρατηρήσεις. Είδαμε πολύ επικοδομητική στάση από αρκετές ομάδες. Βλέπουμε ότι έχουν αναγνωρίσει πως ακολουθούμε μια λογική λύση. Οι σκιώδεις εισηγητές στην πλειονότητά τους ε, νομίζω ότι έχουν τηρήσει αντίστοιχη στάση. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Τελευταία παρατήρηση, κατάθεση τροπολογιών για τις 22 Ιουνίου του 2015, από ό,τι έμαθα, έχει προταθεί να παραταθεί για μία ακόμη εβδομάδα. Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί όντως ήταν πολύ στενά τα περιθώρια. Και δεύτερον, στην τελευταία συνεδρίασή μας με τους κοιόδης ηγητές, είχαμε συμφωνήσει ότι μάλλον θα χρειαστεί να αφιερώσουμε όλο τον, το Σεπτέμβριο για την ε, συζήτηση των, ε, συμβαστικών τροπολογιών για να καταλήξουμε στη ψηφοφορία τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία παρά τις πολυάριθμες τροπολογίες να ε, βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και ένα πόρισμα εργασιών πολύ λογικό. Ευχαριστώ πολύ τον Κνούτ Φλέκνιστον, λέει ο Πρόεδρος. Ακούω τους υπόλοιπους συναδέλφους, έχουν στήσει πολύ το λόγο. Δυστυχώς θα πρέπει και πάλι να σας περιορίσω στα δύο λεπτά τοποθέτησης. Η κυρία Βόζενμπερκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο. Καταρχάς να πούμε ότι ο εισηγητής ο κύριος Φλεκενστάιν έχει κάνει πραγματικά μια πολύ επιμελή προσπάθεια. Μίλησε για μια λογική λύση. Θα έλεγα ότι είναι μια επιμελής και προσεγμένη προσέγγιση. Εκ των πραγμάτων θέλουμε να συμπέσουμε αλλά έχουμε και κάποιες διαφοροποιήσεις. Θα είμαι σύντομη ξεκινώντας από την αναγνώριση ότι αναμφίβολα η διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί προάγει τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία και προπάντων προάγει και τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά στα ζητήματα επένδυση, επενδυτική πολιτική που ενδιαφέρει όλου μα. Κατά την άποψή μα όμω συνδέεται άρρηκτα και με την πρόσβαση στην αγορά. Εκεί έχουμε μια διαφοροποίηση. Νομίζω ότι προϊόν, προϊόντων των προχωρώντας τις διαπραγματεύσεις θα μπορούσαμε να, κάπου να συναντηθούμε. Σε σχέση με τις κοινωνικές διατάξεις που διαπέμπουν το εργασιακό καθεστώς, η άποψή μα είναι ότι αυτέ δεν μπορεί να αποτυπωθούν, να συμπυκνωθούν στον κανονισμό. Είναι απο, ε, αποτέλεσμα διαλόγου, κοινωνικού διαλόγου, σε αυτό συμφωνούμε με την εισήγηση και βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εκεί όπου υπησέρχεται ενδεχομένω μια σύγκρουση με την ε, θεμελιώδη αρχή τη επικουρικότητα. Ε, συμφωνούμε με την εισήγηση ως προς την εξαίρεση της διθοκόρησης και της πλοήγησης σε σχέση με τον κανονισμό. Ως προς τον περιορισμό των παρόχων υπηρεσιών, ε, συμφωνούμε να μπουν κριτήρια. Η διαφοροποίηση στη δική μας την προσέγγιση είναι ότι τα κριτήρια θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα. Να μην έχουν διαφοροποιήσεις που θα μας δημιουργήσουν στην εφαρμογή προβλήματα. Ε, η αφαίρεση τώρα του άρθρου 7 θα πρέπει κατά την άποψή μας να εξετάσουμε κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις διαφάνειας που να σχετίζονται με την επιλογή περιορισμένων παρόχων υπηρεσιών και τούτο, διότι ε, ε, θα είμαι πολύ συντομότατη, δώστε μου μόνο μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, ελοχεύει τον κίνδυνο να μπούμε σε δικαστικές περιπέτειες, να υπάρχουν προσφυγές. Ε, αναφορικά με, του, με τα λιμενικά τέλη, οι λιμενικές αρχές ε, θα πρέπει να τα καθορίζουν αυτόνομα, ότι η αρμοδιότητα στην υποχρέωση δημόσια υπηρεσία που είναι είτε στους φορείς διαχείρισης είτε στην αρμόδια αρχή θα πρέπει ίσως να συμπεριλάβουμε και την άποψη των κρατών μελών. Τελειώνω αμέσως για μια παράμετρο να λάβουμε υπόψη τους μικρότερους λιμένες επειδή έχουν μικρότερο όγκο ως προς τα φορτία μήπως υπάρχει μια δυσανάλογη ε, ε μέτρηση των υποχρεώσεών τους και σε σχέση τελειωτικά για την ε, αυτοτελή ε, διοικητική Αρχή έχουμε την άποψη, ναι κύριε Πρόεδρε είναι ουσιαστικό γι' αυτό το λέω βλέπετε ταχύτατα, η Αυτοτελής Διοικητική Αρχή ε, δεν συμφωνούμε, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εκείνους τους μηχανισμούς ελέγχου μέσα από τους φορείς που διαθέτουν ούτω ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριμένο, ε, στη συγκεκριμένη αποστολή τελειώνοντας να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Φλεκενστάιν, δηλώνουμε αλληλέγγυη στη συνεργασία μας και θα ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος ε, έθεσε. Ευχαριστώ πολύ. Danke sehr. Der nächste ist Peter van Dalen. Gar nicht da? Doch. Voorzitter, dank. Uh, onze steun is op hoofdlijn aan de realistische benadering van de rapport. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συζητή σε σχέση με την οικονομική διαφάνεια. Έχουμε λιμάνια στην Ευρώπη που ξέρουμε ότι χρηματοδοτούνται κρυφά από εθνικές ή τοπικές περιφερειακές αρχές. Δεν υπάρχει διαφάνεια εκεί. Και έτσι δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Για μας η ουσία όλης αυτής της πρότασης είναι η χρηματοοικονομική διαφάνεια. Είναι η γενική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηξίδα για μας, για τις ε, κρατικές επιδοτήσεις δηλαδή. Και γι' αυτό θα ήθελα, επειδή θα κατευθυνθεί στο τέλος του χρόνου, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει τι σκοπεύει να παραγάγει αυτή η Γενική Διεύθυνσή της ε, στο θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σκοπεύω να διατυπώσω τροπολογίες για κάποιες λιμενικές υπηρεσίες, κυρίως εκείνες που έχουν να κάνουν με την πλοήγηση και την πρόσδεση των πλοίων ε, είναι τεράστια σημασία. Δεν πρέπει να κάνουμε οικονομία σε αυτές ε, τις υπηρεσίες ε, και βεβαίως για τις τροπολογίες ξέρω ότι είναι ευρύτατο το πεδίο ε, το νομοθετικό. Πρέπει να αφήσουμε χρόνο να το μελετήσουμε με επάρκεια και γι' αυτό παρακαλώ και πρέπει και εσείς εάν μπορείτε να υποστηρίξετε το αίτημα για την παράταση του χρόνου για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον Κνούτ, τον εισηγητή. Τα κατάφερε όντω να κάνει ένα βήμα περαιτέρω των όσων ε, είχε στην προηγούμενη θητεία το κείμενο. Ε, και να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις. Από τους προαλήσαντες διαπιστώνω ότι είναι καλό να έχουμε περισσότερο χρόνο για τις ε, τροπολογίες. Θα είναι νομίζω, παρά τις πιέσεις που είχαμε μέχρι τώρα τις χρονικές, ε, δυνατόν να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά. Η οικονομική διαφάνεια απόλυτα σημαντική, απόλυτα απαραίτητη. Πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες για τους πάντες. Για το κεφάλαιο 2, πρόσβαση σε αγορές, και οργάνωση, όπως το λέτε τώρα, των ε, λιμενικών υπηρεσιών. Δεν θα έλεγα ότι είναι ε, στρεβλή αλλαγή, ότι θα διαστρεβλώνει την εικόνα αυτή η αλλαγή του τίτλου, αλλά εν περιπτώσει θα ήθελα κάπου να βλέπω αυτή την ιδέα ότι πρόκειται για πρόσβαση στις αγορές. Και όταν ε, μιλάμε για Αγγλία όπου είναι ιδιωτικές, ιδιωτικοί λιμένες, όταν μιλούμε για άλλες περιοχές ή κράτη που έχουν δημόσιους λιμένες, αλλά οι λίμενοι εργάτε μπορεί να εργάζονται ως ιδιώτες και όλα αυτά είναι συνθήκε τι οποίε θα πρέπει να εξετάσουμε και να ε, ε, μελετήσουμε. Επίσης θέλω να δω εάν υπάρχει μία προσφορά για εξαγορά ε, ενό τομέα υπηρεσιών, εάν στην προσφορά αυτά περιλαμβάνεται, θα πρέπει να δηλώνεται αν περιλαμβάνεται και η ανάληψη των εργαζομένων στην ομάδα του ε, αγοραστή. Στις συνθήκες ε, παραχώρησης πρέπει να κοιτάξουμε επακριβώς τι ε, προβλέπεται για τους λιμένες. Στο κεφάλαιο 4 παραδείγματι όπου λέει το Συμβούλιο ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες οι λιμενικές να είναι πάντοτε προσβάσιμες δημόσια για όλους τους χρήστες για όλους και όλες οι υπηρεσίες, δηλαδή να μην γίνεται το cherry picking, να μην διαλέγει κανείς ότι θα πάρει τη μία ή την άλλη υπηρεσία μόνο. Για δε την εποπτική αρχή, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιπλοκό, το Συμβούλιο έχει πολύ καλύτερη πρόταση και γι' αυτό νομίζω ε, ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε πως και ο εισηγητής αλλά και το Συμβούλιο έχουν δείξει πολύ πιο ρεαλιστική και πρακτική στάση στην υπόθεση αυτή. Thank you, Mr. President. Εμείς καλωσορίζουμε τις, ε, καλωσορίζουμε θετικές αλλαγές που περιέχει το... η πρόταση, η έκθεση του κυρίου Φλίκεστάιν. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα... την απομάκρυση της ε, πρόσβασης των αγορών μέσα στο κείμενο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στους τελευταίους τρεις μήνες ε, είχαμε τρεις θανάτους στα ευρωπαϊκά λιμάνια εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευση και επαρκών μέτρων ε, ασφαλείας. Γι' αυτό λοιπόν στην ΚΟΕ, ως ΚΟΕ υποστηρίζουμε πλήρως την ε, εισαγωγή τροποποιήσεων του κυρίου Φλίνκεσταϊν που αφορούν την, ε, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον κοινωνικό διάλογο και τα δικαιώματα των εργατών. Είμαστε απολύτως υπέρ της διαφάνειας σε όλους τους τομείς. Απλώς δεν πρέπει η διαφάνεια να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσχημα ε, για, την, ε, για να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα αφαιρέσουν δικαιώματα από τους εργαζόμενους καθώς επίσης και θα μειώσουν τα μέτρα ασφαλείας. Και είμαστε επίσης έτοιμοι να δουλέψουμε με το Κοινοβούλιο και με τον κύριο Φραγκεστάιν στη συνέχεια για να ε, αναπτύξουμε ε, και να τροποποιήσουμε προς το καλύτερο την πρότασή του. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Φράγκενστάιν, σας ευχαριστούμε για τη δουλειά σας όσο κάνατε μέχρι τώρα. Τρίτη προσπάθεια και καλύτερη. Να επαναλάβω αυτό το οποίο προανέφερα όσον αφορά το ότι χρειάζεται διαφάνεια στη μοτοδότηση την κρατική. Δεν είναι δυνατόν να φροντίσουμε τα λιμάνια χωρίς να υπάρχει χρήμα κρατικό για την υποδομή, για τη λειτουργία και όπως προείπα έχουμε ιδιωτικοποίηση σε όλα τα λιμάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, βέβαια εδώ μιλάμε για την Ευρώπη. Μ' αρέσει η πρωτοβουλία κύριε Φλέκεστάιν του να κάνουμε τη Γενική Διεύθυνση την Αρμόδια μια συνάντηση για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι ε, κρατικέ ενισχύσει. Ε, συμφωνηθεί κάτι κάποια στιγμή. Δεν έχει νόημα το να προχωρήσουμε βιαστικά για αυτόν τον κανονισμό. Επομένω, να έχουμε ένα τουλάχιστον σχέδιο κειμένου για αυτέ τι κρατικέ βοήθειε. Επίση, είναι πολύ σημαντικό κάθε νομοθετικό πλαίσιο να σέβεται την πολυμορφία, την ποικιλία που υπάρχει στην Ευρώπη όσον αφορά τα λιμάνια. Από πλευρά γεωγραφική, από πλευρά μεγέθου, οργάνωση, ε, διαχείριση, τι αγορά εξυπηρετεί το κάθε λιμάνι. Και σε σχέση με αυτό, κύριε Φλέγκενστάιν, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ενιαία, μοναδική μέθοδο για όλους. Άρα ε, γι' αυτό και πιστεύω ότι από το κεφάλαιο 2 τα σχετικά με την πρόσβαση θα πρέπει να διαγραφούν. Έχω σημειώσει εδώ ένα σώρο και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που είπατε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για κοινωνικέ ε, διατάξεις, να μην έχουμε την εκμετάλλευση των ε, εποχιακών και προσωρινών εργαζομένων, Επίσης ε, τα σχετικά με τις βυθοκόρους θα πρέπει να τα επαλείψετε από τον κανονισμό. Και εγκατακλείδη έχω να σας πω το ότι εμείς σαν στόχο έχουμε αυτή η πολιτική να ενταχθεί στο στόχο μας για βιώσιμες μεταφορές, σεβόμενοι το περιβάλλον, σεβόμενοι τους χρήστες, με το μάτι στο μέλλον. Η κυρία Δαμάτα. Oh, Πίτερ Lundgren. Και ο Πέτερ Λούντκριν. Σας ευχαριστώ. Α, μα δεν έχετε εγγραφεί ως ε, ομιλήτρια, τέλος πάντων. Μα είμαι σκιώδης όμως, λέει η κυρία Δαμάτα. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Παρά το ότι το Πρόεδρο της Επιτροπής θέλει να ανοίξει την αγορά όσον αφορά τον ανταγωνισμό και έτσι να σταματήσουν τα μονοπόλια. Όμως, όμως, κάποια σημεία αυτού του χανισμού, ιδίως όταν τα μικρά λιμάνια δημιουργούν προβλήματα. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης όσον αφορά τα λιμάνια στον Βορρά. Βεβαίως υπάρχει περισσότερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη, πιο αποτελεσματική διαχείριση, πιο εύκολη. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτή η διάσταση μεταξύ Βορρά και Νότου και επομένως ε, δεν μπορούμε να έχουμε τι ίδιε προϋποθέσεις, τα ίδια πρότυπα για να έχουμε ε, μια αποτελεσματικότητα και για να δούμε πώς θα ανοίξουν οι υπηρεσίες. Έτσι αυτός ο κανονισμός ε, είναι φτιαγμένος για το βορρά. Και λέει όντω ότι η γραφειοκρατία δεν κάνει καλό στην αποδοτικότητα, στην οικονομία, χαχυροτερεύει τι υπηρεσίε. Δεν θα πρέπει επομένως τα μικρά λιμάνια να τα επιβαρύνουμε με ένα πλαίσιο δυσανάλογα μπλεγμένο. Και επομένως θα πρέπει να δούμε το ότι το να υπάρχουν πάρα πολλοί που παρέχουν τις υπηρεσίες δεν βοηθάει. Υπάρχει ανταγωνισμός, ε, θα πρέπει να σεβαστούμε και το περιβάλλον, οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε ε, πάρα πολλούς παρόχους υπηρεσιών και αυτό θα πρέπει να κρυθεί κατά περίπτωση. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στα ευρωπαϊκά λιμάνια και διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης. Και αυτό μας ανησυχεί ότι δεν ελήφθη υπόψη. Αυτή η ποικιλομορφία, οι διαφορές. Επίσης, πρόκειται να ζημιωθούν από αυτές τις ρυθμίσεις τα λιμάνια της Μεσογείου. Να δούμε τι γίνεται και με τα κοινωνικά θέματα, τι γίνονται με διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων ας πούμε αυτό που λέει η συγγήτρια, ε, ο εισηγητής μάλλον για την ε, μετάθεση, μεταφορά ε, του προσωπικού. Ας πούμε όταν έχουμε κάποιο διαγωνισμό, κάποιες προμήθειες, θα πρέπει να δούμε πώς θα κατοχυρώνονται από τέτοιες κινήσεις οι θέσεις των εργαζομένων. Αυτό αφορά και τους πλοηγούς που και αυτό είναι μια οικονομική υπηρεσία. Να δούμε τι θα γίνει με τον παράγοντα διαφάνεια σε κάθε περίπτωση επένδυσης κρατικών πόρων θα πρέπει να είναι δεδομένη, αυτονόητη η διαφάνεια. Θα πρέπει επομένω ε, αυτό να το ελέγξει και το ελεγκτικό συνέδριο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά... πέραν το τη ε, ανάγκη εναρμόνιση να αφήσουμε περιθώριο ελεγμό στα κράτη-μέλη και στι λιμενικές αρχέ. Χρειάζεται... Ναι, αλλά τώρα πρέπει να διακόψω. Ε, όχι, όχι, πρέπει να διακόψω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλά δεν θα ήταν δίκαιο για, για τους λοιπούς. Κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή ο οποίος πραγματικά δυσκολεύτηκε. Ο Πίτερ είναι εισηγητής της ομάδας ECR και ναι, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδιωτικοποίησαμε τα λιμάνια πριν 30 χρόνια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη ε, εισήγηση έτσι ώστε να μην έχουμε αρνητικέ επιπτώσεις. Έχουμε περιθώρια λιγμών, έχουν γίνει πολλοί συμβιβασμοί. Νομίζω ότι για τις προσδέσεις και για τα καύσιμα των πλοίων έχουμε κάποια ζητήματα και χαίρομαι πως ε, ε, τουλάχιστον για το θέμα των πλοηγών υπάρχει αναγνώριση από πλευρά του εισηγητή για το τι συμβαίνει. Και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, για παράδειγμα ε, χρήση του εργατικού δυναμικού. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, καταργήσαμε ε, το Σωματείο των Αχθοφόρων όπου πραγματικά οι συνθήκες εργασίες ήταν φρικτές. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να τα ξανασκεφτούμε τα θέματα αυτά μία παρέκκληση για τα μικρά λιμάνια φαίνεται να εξαφανίστηκε και δεν βλέπουμε την παρέκκληση αυτή που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να παραμείνει στο κείμενο διαφορετικά κινδυνεύουν τα λιμάνια αυτά και για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, τα PSO, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να επιβληθεί αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να διακρίνουμε. σας ευχαριστώ πολύ. Και που το χρόνο ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συμφωνώ με του προελίσσαντες συναδέλφου, ότι η έκθεση Φλέκεστάιν η δεύτερη έκθεση αυτού θα μας βοηθήσει πολύ. Η προσέγγιση του εισηγητή είναι πρακτική, είναι ρεαλιστική Τώρα θα προχωρήσουμε στο θέμα της ε, απορρίθμιση για του λιμένε. Αλλά ερωτώ, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια στα οικονομικά και πώς θα εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα. Γιατί θα πρέπει το ένα να προηγηθεί και κατόπιν θα δούμε τι ισχύει με το δεύτερο. Πώς θα προχωρήσουν αυτά τα δύο ζητήματα χέρι-χέρι, πώς θα δούμε στην πράξη τι ισχύει. Τώρα όσον αφορά τις λιμενικές υπηρεσίες και τους αυτών των υπηρεσιών, δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν το cherry picking την επιλογή. Θα πρέπει οι λιμενικές αρχές να είναι θέση να πούν ότι κανείς όταν σε ένα λιμάνι θα πρέπει να ε, γίνεται μέτοχος όλων των υπηρεσιών και όχι ορισμένων του λιμάνιου. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ε, αμοιβόμενους με ημερομίσθιο. Ε, αυτό είναι πολύ ψευδρομικό σύστημα γιατί στην αγορά εργασία υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια ρύθμιση πιο ευέλικτη. Μάλιστα. θέλετε. Α, ο Ιβο συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τον εισηγητή για την εκθέσή του και να κάνω μερικέ παρατηρήσει που ακούσαμε και από την κυρία Βόζεμπερ και από τον κύριο Φαντεν Κάμπ. Ο εισηγητή λέει ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, κανένα insights μοντέλο. Αυτό είναι αλήθεια, συμφωνούμε κι εμεί. Υπάρχουν λιμένε με διαφορετικά πρότυπα διαχείριση στα κράτη-μέλη, πάλι μάλιστα ορισμένα εκ των οποίων πρόσφατα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και του δεν υπάρχει λόγο να μην διαφυλαχθούν αυτά τα πρότυπα διαχείριση αφού τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώς τηρούν τους κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά και τις ε, χρηματοοικονομικές, την χρηματοοικονομική διαφάνεια. Για το PSO, Public Service Obligations, υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ε, το cherry picking που ακούστηκε νωρίτερα, προφανώς και ισχύει και για τους λιμένες, Πρέπει να υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, της λιμενικές. Μπορεί να χρειαστεί να επιβληθεί αυτός ο κανόνας της ε, παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ακριβώς για να μην προσπαθήσει κάποιος φορέας εκμετάλλευσης να επιλέξει με το cherry picking αυτές τις υπηρεσίες που τον βολεύουν. Επίσης ε, εδώ θα θέλαμε να μπει το κομμάτι αυτό όχι μόνο σε θεολογική σκέψη αλλά και σε, στο διατακτικό του κειμένου. Θα κάνουμε τη σχετική τροπολογία και κάποιες άλλες παρατηρήσεις που ακούστηκαν κύριε Πρόεδρε, η πλοήγηση, όπου συμφωνούμε πως είναι η υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να μείνει εκτός του πεδίου και το ίδιο και για τη βυθοκόρηση. Να αποκλειστεί δηλαδή από την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρκος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά σε ένα πολύ δύσκολο τομέα. Ε, πολύ επιγραμματικά μόνο και μόνο και από την ελληνική πλευρά για να δείξουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Ε, πρώτο, ευαισθησία στην άσκηση τιμολογιακής πολιτικής. Φανταστείτε μια χώρα που είναι σε ε, τόσο έντονη οικονομική κρίση και ταυτόχρονα έχει έναν επίσης έντονο ανταγωνισμό που λιμάνια εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές έχουν και κρατική επιχορήγηση. Ε, το δεύτερο είναι το θέμα της οικονομικής διαφάνειας, φυσικά το στηρίζουμε 100% αλλά να προσθέσουμε την ανάγκη να εξαιρεθούν οι μικροί λιμένες από την παράγραφο 2 του άρθρου 12 σχετικά με την τήρηση χωριστών λογαριασμών γιατί σε ένα μικρό λιμάνι με μικρό ε, φορτίο το διοικητικό κόστος είναι δυσανάλογο, όχι βέβαια εις βάρος της διαφάνειας. Ε, τρίτο αυτό που λέμε για τη διαφάνεια των διαβουλεύσεων με τους χρήστες του λιμένα, αυτό εμείς στα ελληνικά λιμάνια γίνεται σε αρκετό βαθμό, ε, λέμε λοιπόν ναι στην ανάγκη διαβούλευσης, όχι όμως σε ένα δεσμευτικό χαρακτήρα αυτήν. Και τελειώνοντα, θεωρώ πω η πρόταση βελτιώνει την απόδοση του λιμένου και δίνει την πρέπουσα σημασία στη διαφάνεια που δημιουργεί συνθήκε την προσέλκυση επενδύσεων. Ευχαριστώ πάλι τον, επενδύτη, τον ε, εισηγητή. Danke sehr, jetzt τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η μεγάλη διαφορά σε σύστημα και σε μεγέθη λιμενών και οι παλαιές παραδόσεις στις βίες κοινωνικής ε, συγκρούσεις που είχαμε είναι ένα κομμάτι από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είναι η τέταρτη ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξέρετε πως έχουμε περάσει πολλά θερμά επεισόδια εδώ τα περασμένα χρόνια. Πολύ καλή έκθεση, πολύ δουλεμένη ε, πολλές από τις θέσεις ε, για την ευελιξία, για το διοικητικό βάρος ε, τα κτλ. Ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Ε, πλοήγηση, ναι, πάει στο θέμα αυτό. Είμαι συγχωρείτε πλοήγη. Κοιτάξτε, υπάρχει διαφορά μεταξύ λιμενικής αρχής και λιμενικού ταμείου. Για κάποιες χώρες είναι το ίδιο, και κάποιες δεν είναι και είναι δύσκολο να τα βάλουμε αυτά στο ίδιο καλάθι. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχές αυτές να μην ασχολούνται με την διαχείριση. Γιατί αν οι αρχές επιβάλλουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο διαχειριστή, θα πρέπει ο διαχειριστής να έχει και την ευθύνη να παρακολουθεί τις συναλλαγές στο λιμάνι, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πολλές δυσκολίες, για παράδειγμα σε ιδιωτικά λιμάνια που δεν έχουν λιμενική αρχή για να το πω έτσι. Και έχουμε και κάποιε άλλε που δεν έχουν λιμενική αρχή, αλλά λιμενικό ταμείο. Έχουμε λοιπόν αυτή την επιφύλαξη. Αν ο έλεγχο είναι τελείω διαφορετικό, ανάλογα με το ε, σε ποιο κράτο μέλο βρίσκεσαι, τότε θα αντιμετωπίσουμε πραγματικέ δυσκολίε για να κάνουμε ελέγχου οι οποίοι θα είναι και αποτελεσματικοί αλλά και συγκρίσιμοι. Άρα λοιπόν αντίθετα με τον εισηγητή πιστεύω εδώ, και εδώ είναι το μεγάλο σημείο στο οποίο ε, διαφωνώ μαζί του, δεν γίνεται δεν γίνεται να μην κάνουμε τέτοιου ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κοινό τρόπο, γιατί διαφορετικά κάποιοι δεν θα ελέγχονται. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ έχει το λόγο μετά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμμετείχα σε τουλάχιστον τέσσερις προτάσεις και χαιρετίζω αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Ας πίσω να καρποφορήσει περισσότερο από προηγούμενες φορές. Ε, να σας πω πως εγώ είμαι μάλλον υπέρ. Αν πρόκειται να το αδειάσουμε από οποιαδήποτε ε, τεχνική λεπτομέρεια, ας το αφήσουμε ησυχό, αλλά εν πάση περιπτώσει η νέα πρόταση που κάνετε είναι ενδιαφέρουσα. Παρόλο που επαναλαμβάνει κάποια θέματα, ό,τι έχει να κάνει με την ε, εξυγίανση, με την ενίσχυση, με τον κοινωνικό διάλογο, μια χαρά αλλά αυτό το κάνουμε και σε άλλους κλάδους. Χαίρομαι που τα έχετε εδώ, χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και κάποια άλλα ε, στοιχεία στο κείμενο. Να δούμε βέβαια το Συμβούλιο σε ποιο βαθμό θα τα δεχτεί. Μιλάμε για κρατικές ενισχύσεις. Να τοποθετήσουμε αυτό σε ένα εκτιμώντας, κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν διαυκολύνει την ε, διαφάνεια. Εμεί πάντα λέγαμε πως αυτό που χρειαζόμαστε είναι όχι ανταγωνισμό μεταξύ λιμένων, αλλά διαφάνεια. Και επιτέλους κάποιος αναγνώρισε πως υπάρχει μια εδώ δημόσια υπηρεσία που πρέπει να προσφέρεται, αλλά θα πρέπει να έχουμε διαφάνεια και ανταγωνισμό μεταξύ λιμένων επί ίσης ώρες. Δεν ξέρω αν τα σχετικά άστρα, το 14 για παράδειγμα και το 2015 βελτιώνουν τη διαφάνεια ή αν απλώς λέμε εντάξει ας συνεχίσουμε όσο έχει κατάσταση αφού σε κάποιο βαθμό έχουμε διαφάνεια. Ας βελτιώσουμε λοιπόν τις επιδόσεις μας εκεί. Και τέλος είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου η αν απλω λεμε ενταξει που έκανε ο ας βελτιωσουμε λοιπον τι επιδοσει μας εκει και ότι αποφασίζει η Μαδρίτη τι κάνουν στη Βαρκελόνη. Δεν το αποφασίζει η Μαδρίτη, το Ισπανικό Κοινοβούλιο το αποφασίζει. Το ίδιο κάνει και το Bundestag στη Γερμανία, κύριε Σιγητά. Εντάξει, στο κάτω-κάτω μην μου πείτε πως ε, μπορούμε να πούμε εδώ για παράδειγμα πω το Βερολίνο αποφασίζει τι συντάξει θα παίρνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πολύ φυσιολογικό το Ισπανικό κράτος να αποφασίζει τι λιμενικά τέλη θα επιβάλλει στους λιμένες όλους τη χώρα. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Λούση Άντερσεν. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω έκανε πολύ τολμηρή προσπάθεια ο εισηγητή, τόσο ώστε να παραμείνει στο θεματολόγιο της έκθεσης το θέμα της κρατικής βοήθειας ως και αν δεν του ήταν εύκολο και επίσης ε, λάβουμε πως αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι το ότι θα πρέπει ο κοινωνικός διάλογος θα δημιουργεί εργαζόμενο όλα αυτά να καλυφθούν να καλυφθούν και να προβληθούν πολύ σημαντικά και για μας παρ' όλα αυτά άκουσα και είπε η Τζάκη πριν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε τελείω διαφορετική κατάσταση από ότι τα άλλα ε, κράτη-μέλη σε σχέση με αυτό ε, αυτό ισχύει για τα συνδικάτα εκεί, για τα βασικά λιμάνια. Οπότε θα προτιμούσαμε εμεί να μην υπάρχει καθόλου μια ρύθμιση από αυτού. Επίση, λαμβάνω υπόψη αυτό το οποίο είπε και ο Κίθ σε σχέση ιδίω με το κατά πόσον βιαζόμαστε να κλείσουμε στο γόνατο αυτό το κείμενο. Γιατί θέλουμε ε, γενικότερη το, το τοπίο να αλλάξει ιδίω όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ρύθμιση για τα λιμάνια που τελικά να βοηθάει και την απασχόληση ε, και την ανάπτυξη και τη δικτύωση. Και ήθελα να σας πω ότι πώς είναι εδώ να έχουμε καλύτερη νομοθεσία για οι Έχουμε και το κείμενο των ε, θεσμικών οργάνων για την καλύτερη νομοθεσία ή κοιτάξτε τι λέει η κοιτάξτε τι λέει η Κομισιόν, τι λέει το Συμβούλιο, τι κάνουμε εμείς. Κάνουμε αυτά που λέει αυτό το θεσμικό κείμενο. Υπάρχει έτσι νομίζω ότι κανονισμός. Έχουμε όμως τώρα το καινούργιο σχέδιο κειμένο. Και νομίζω ότι εάν θέλουμε να αλλάξει σημαντικά το καθεστώς, θα πρέπει πρώτα να έχουμε μια μελέτη επιπτώσεων και για την οικονομία και για το περιβάλλον. Πού είναι αυτή η μελέτη? Δεν ναι, καθυστέρησε εδώ να το βρούμε. Να, να σα πω μία παράγραφο από αυτό που λέει το κείμενο. Λέει ότι η συμφωνία θέσεων οργάνων θα πρέπει η νομοθεσία να είναι σφαιρική, να είναι ξεκάθαρη και να μπορούν πολίτε να, να ξέρουν δικαιώματα και υποχρεώσει. Επίση και να υπάρχουν και ε, οι μελέτε των επιπτώσεων και να μην έχουμε δυσανάλογο κόστο. Ε, είναι εδώ να, να είναι εφαρμόσιμα τα όσα νομοθετούμε. Και οπότε, για πέστε με εδώ πέρα, θεωρείτε ότι το κείμενο συμμορφώνεται προ αυτά Πάρα πολύ καλά τα, τα προσπάθησε ο εισηγητής, αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό που σας διάβασα. Ευχαριστώ. Πίτερ Λούγκρεν. Πρόκειται για πρόταση που αφορούσε την πρόσβαση στις αγορές. Να δούμε τι περιορισμού θέλουμε να θέσουμε για να πετύχουμε το στόχο μα. Εγώ συμφωνώ στα όσα λέτε για την διαφάνεια, αλλά είναι σημαντικό επίση αυτοί που χρησιμοποιούν του λιμένε να είναι δυνατόν να έχουν συμμετάσχει σε κάποια διαβούλευση για αυτό το νομοθέτημα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτού να ρωτήσουμε, αυτού που προσφέρουν τι σχετικέ υπηρεσίε, ε, ούτω ώστε να υπάρχει περιβάλλον εργασίας ε, αξιοπρεπέ, να υπάρχει κατάρτιση, ε, γιατί μιλάμε τώρα για δουλειά με πάρα πολύ βαριά μηχανήματα. Και έτσι τελικά να μειώσουμε τα ατυχήματα στο χώρο εργασία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομο. Σοφόντο, το και τώρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σα. Θα είμαι κι εγώ σύντομο. Δεν θα σας περιγράψω όλες τις στοιχείες της ε, μελέτης αξιολόγησης στις οποίες στηρίχθηκε αυτή η τόσο σημαντική έκθεση μια μελέτη αξιολόγηση που ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε έρθει εδώ για τρίτη φορά με ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα θα καταγράψω το πόσο πυκνά ήταν τα σχόλιά σας και οι διάφορες παρεμβάσεις σας Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και την έκθεση Φλάνκενστάιν νούμερο 2. Για την διαφάνεια είναι μια βασική συνεισφορά την οποία πραγματικά χρειαζόμαστε για να διευκολύνουμε την παραγωγή και την έγκριση ε, κάποιων μαζικών εξαιρέσεων που να καλύπτουν ε, λιμάνια ε, και μία μαζική εξαίρεση η οποία είναι λογική που δεν λαμβάνει υπόψη μόνο το ύψος των επενδύσεων Άρα και άλλες παραμέτρους. Είναι πολύ σημαντικό. Χαιρετίζουμε επίσης την επιπλέον σημασία που δίνεται στην αυτονομία και κυρίως στην οικονομική αυτονομία των λιμένων. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να διακρίνει κανείς ε, τις διαφορές μεταξύ των διαχειριστικών φορέων των λιμένων και των λιμενικών αρχών. Επίσης, η κοινωνική διάσταση αυτής της έκθεσης, κάποιες από που ακούστηκαν ήταν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Uh, when uh, uh, at... Θα τα δούμε όλα πολύ προσωπικά. Για παράδειγμα, για τους αχθοφόρους. Λόγω της περασμένης προϊστορίας αυτού του φακέλου είπαμε να μην το συμπεριλάβουμε στην πρόταση. Κάτι ακόμα η υποχρεωτική μεταφορά δικαιωμάτων δεδομένων των τόσο διαφορετικών καταστάσεων όπως να κράτη-μέλη, όπως επίσης και της ε, μεταλλασσόμενης εργασιακής αγοράς που στην οποία αναφέρθηκαν τουλάχιστον δύο ομιλητές σήμερα, είπαμε στο σημείο αυτό να κινηθούμε προσεκτικά για τις υπηρεσίες, λιμενικές υπηρεσίες. Χαιρόμαστε που ο εισηγητής προσπαθεί να διευρύνει την έννοια, ακόμα και ο τίτλος έχει αλλάξει για να φανεί αυτό μιλάμε για διαφορετικά στοιχεία για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και νομίζουμε ότι εδώ θα πρέπει να διατηρήσουμε την αρχή της επιλογής. Σας παροτρύνω λοιπόν να συνεχίσετε να στηρίζετε ένα κείμενο το οποίο ξεκαθαρίζει πως η αρχή της επιλογής είναι η βασική αρχή έτσι ώστε να διευκολύνουμε και το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητό. Κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε εδώ είναι μια κωδικοποίηση των διαδικασιών ε, για την επιλογή των λιμενικών υπηρεσιών. Γιατί? Για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Για να αποφύγουμε καταγγελίες και ενστάσεις που κοστίζουν ακριβά σε όσους διαχειρίζονται λιμάνια. Και τέλος, για να εκτιμήσουμε εμείς καλύτερα το πώς γίνονται οι έλεγχοι, αλλά και το τι συμβαίνει όταν τον έλεγχο του λιμανιού αναλαμβάνουν επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει δηλαδή αυτές οι επενδυτικές αποφάσεις να ελέγχονται μέσω κάποιου είδους κωδικοποιημένης διαδικασίας αυτό που προτείναμε εμείς ήταν κάπως μακροσκελές ήταν δηλαδή κάτι παρόμοιο με αυτό του δικαιώματος εκχώρησης ε, είπε να συνοψίσει τον κατάλογο το Συμβούλιο ίσως εδώ υπάρχει χώρος για να βελτιώσουμε τα πράγματα τώρα για την πλοήγηση γιατί θέλετε να το βγάλουμε Είπαμε πάντα πως μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα γιατί λοιπόν να μην έχουμε αποκλειστικό δικαίωμα και για τους πλοηγούς στα λιμάνια. Με γενικές διαδικασίες με δικαίωμα επιλογής. Και τέλος για το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Εμείς με ευαισθησία αντιμετωπίζουμε κάποιες από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Θα μπορούσαμε να εξαιρέσουμε τα μικρά λιμάνια και με συμπάθεια αντιμετωπίζω τα επιχειρήματα που ακούστηκαν. Ο κανονισμός όντως ουσιαστικά αναφέρεται σε λιμάνια με ευρωπαϊκά μεγέθη δραστηριότητας. Έχουμε τις κατευθύνσεις γραμμίες για τα τέντη, οπότε ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι τα λιμάνια αυτά που συμπεριλαμβάνονται. Αυτό να είναι το βασικό πλέγμα λιμένων και ίσως το επίπεδο αυτό που έχουμε στα τέντη να είναι το σωστό για να καλύψουμε. Ευχαριστώ πολύ ο εισηγητής να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επισέλθω σε όλες τις παρατηρήσεις. Πολλά θα χρειαστεί να συζητήσουμε και στο πλαίσιο της ε, αντιπαράθεσης ε, με τις ε, τροπολογίες. Αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα στήματα ώστε να έχει γίνει παρεξήγηση και να κάνω και μερικές παρατηρήσεις. Καταρχάς για την κυρία Γιάλα Σέντερ. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για τους φόρους, αλλά για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης για τον λιμένα. Ούτε στη Γερμανία τα ορίζει το Bundestag. Το Αμβούργο, Φερρυπίν, έχει προφανώς αντισταθεί πολύ. Αλλά μπορούμε να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει. Δεύτερον, ξέρω ότι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα οι λιμένες στη Βρετανία. Και τον τελευταίο γύρο συζητήσεων είχα πει ότι η Βρετανία θα συμφωνούσε με μία φράση «Χρήματα για όλους τους λιμένους που δεν, δεν βρίσκονται σε νησί». Αλλά, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με αντικειμενικά προβλήματα. Αντικειμενικά προβλήματα λοιπόν πρέπει να τα δούμε με σοβαρότητα. Είχα πάει και στο Λονδίνο και θα ήθελα να πω γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα. Πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν σαν επικρίσεις είναι αισθήματα που με είχαν απασχολήσει και εμένα και είχα πει στον εαυτό μου, μα και εσύ αυτό θες. Τι θα κάνουμε με τους πιο μικρούς λιμένες Φερρυπίν. Πρόσβαση διαφορετική στις αγορές. Γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες. Ναι, και εγώ αυτό θέλω. Άρα λοιπόν μπορεί να μην έχω βρει την κατάλληλη διατύπωση σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι νοητή μια διαφορετική, καλύτερη διατύπωση που μπορεί να προκύψει μέσα από τη συζήτηση και πολλές φορές να τη δεχτώ. Διαφάνεια και προσβάσεις αγορές νομίζω ότι μπορούν να συγκεραστούν. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κόστος, αλλά με διαφάνεια των κριτηρίων για να ξέρουμε πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια. Να μην είναι αυθαίρετος ο προσδορισμός για το cherry picking, το ξεδιάλεγμα βεβαίως. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ εύστοχο το επιχείρημα και το έχω συμπεριλάβει και εγώ. Εάν τυχόν η διατύπωσή μου δεν σας ικανοποιεί θα βρούμε μια καλύτερη. Επίσης, παρατηρήσεις τώρα. Μπορεί να λέμε ότι κάποιες διατάξει μπορεί να είναι πιο πρόσφορες για λιμένες του βορρά, από ό,τι για του Νότου, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας κλπ. Ωραία. Αλλά αν είναι έτσι, αν έχετε δίκιο, τότε θα κοιτούσα να αλλάξω τις διατάξεις που αφορούν τους βόρειους λιμένες και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστούν με κάποιες τροποποιήσεις αυτά στους λιμένες του Νότου, χωρίς βέβαια να προκύψουν ιδιαίτερε δυσκολίες ή προβλήματα. Η αγορά εργασίας αλλάζει, λέτε. Και βεβαίω πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό. Αλλά επανέρχομαι για να πω το εξή. Εάν πρόκειται να διατυπώσουμε διαφορετικά το κείμενο, θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε να μην τροποποιήσουμε όσο και αν αναφερθούμε ενδεχομένω στέλνοντα ένα μήνυμα στι εργασιακέ σχέσει δεν μπορούμε μόνο να τι διαταράξουμε όπω έχουν διαμορφωθεί γενικά οι εργασιακέ σχέσει στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να έχουμε καλέ εργασιακέ σχέσει κτλ. Με μία φράση, με ένα μήνυμα, με μία αρχή επικουρικότητα, με οποιοδήποτε κριτήριο που μιλάει για κοινωνικό διάλογο, όπου έχουμε αρμοδιότητα. Και όποιο έχει αρμοδιότητα, γιατί δεν έχουμε εμεί την αρμοδιότητα να ορίσουμε αυτέ τι ε, διατάξει. Ώστε όταν πηγαίνει κάποιο να δουλέψει ένα λιμάνι, να ξέρουμε ότι μπορεί να μην αλλάξουμε τις εργασιακές συνθήκες όπως γενικά επικρατούν στην Ευρώπη, αλλά πάντως δεν θα επιτρέψουμε επιδείνωσή τους ειδικά στους λιμένες. Για δε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και την πρότασή της για τις κρατικές ενισχύσεις. Εάν θεωρείτε ότι δεν σας αρκούν οι προτάσεις αυτές, έχετε βεβαίω κάθε δυνατότητα στην ψηφοφορία να εκδηλώσετε την αντίθεσή της. Είπαμε ότι είμαστε, γιατί σημαίνει να κάνουμε όσο δυνατόν πιο πολλούς συμβασμούς ε, και αυτό θα το δούμε όταν και στους δύο τομείς έχουμε προχωρήσει αρκετά στο να δούμε προς τα που κλείνει η πλάστιγκα. Διαφορετικά μπορεί με το ένα χέρι να δίνουμε αυτό που παίρνουμε από το άλλο. Για το Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι είναι καλό από τις προτάσεις του Συμβουλίου, από τις θέσεις του Συμβουλίου και τι μπορούμε να κρατήσουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε και διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε έναν συμβιβασμό ο οποίος δεν θα είναι πάντα απόλυτα ικανοποιητικός. Θα πρέπει να κοιτάξουμε από όσα έχει κάνει δεκτά το Συμβούλιο τι μπορούμε να αντέξουμε κι εμείς και να βρούμε τη χρυσή τομή. Δεν είναι δυνατόν όμως από την άλλη να αντιγράφουμε οτιδήποτε έχει δεχθεί το Συμβούλιο. Παραδόξω πω δεύτερη φορά και κατ' το Συμβούλιο έχει δουλέψει πιο νωρί από εμά. Είναι ταχύτερο, αντέδρασε πιο νωρί από ότι εμείς. Ας το δούμε και αυτό. Κάθε πράγμα στον καιρό του, αλλά όσο το δυνατόν ό,τι κάνουμε το κάνουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κνούτ Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ όλου όσοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Τροπολογίε μια και το ζητήσατε, παραδένουμε την προθεσμία 29 Ιουνίου τώρα, η προθεσμία για τις τροπολογίες, 29 στη μεσημέρι. Το επόμενο θέμα και κλεισμένο των θυρών. Οι συγκητές τριμερούς διαλόγου. Ούτε η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να μείνει.